η βελτίωση της υγείας των μητέρων, να μειωθεί η θνησιμότητα των παιδιών και τα ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σε ορισμένες χώρες η θέση των γυναικών έχει επιδεινωθεί. Γι' αυτό και είναι οι γυναίκες πάντα στα χέρια των ανδρών, δηλαδή του πατέρα τους, του συζύγου, των αδερφών και είναι κρίμα που χρησιμοποιούν τη τεχνολογία εχμής για να προγραμματίσουν την σύνθεση της οικογένειας. Οι γυναίκες επιλέγουν να έχουν λιγότερα παιδιά εξαιτίας των οικονομικών εξελίξεων και τα μωρά θερούνται πολλές φορές βάρος. Τώρα η πρακτική που γίνεται για την επιλογή του φίλου κατά τη γέννηση έχει σαν αποτέλεσμα να γεννιούνται περισσότερα παιδιά και οδηγεί σε μια κοινωνική συμπεριφορά η οποία ενισχύει τη βία, την αστάθεια, την ανασφάλεια, αλλά έχει και αρνητικές επιπτώσεις στην γονιμότητα και τελικά σε εθνισμότητα των αντινάμει ε, μητέρων. Πρέπει να μελετήσουμε βέβαια βαθύτερα τις αιτίες και να αναλύσουμε τι οικονομικά κίνητρα υπάρχουν που οδηγούν σε τέτοιες πρακτικές και αυτό το στηρίζω με τις τροπολογίες μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει τη βελτίωση της εκπαίδευσης, να υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τις γυναίκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί με τις ε, εθνικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές για να ενισχυθεί μια τέτοια πολιτική υπέρ των γυναικών και να καταργηθούν οι πρακτικές αυτές. Επίσης, πρέπει να κοιτάξουμε και την ενίσχυση της νομοθεσίας όσον αφορά την βία κατά των γυναικών, αλλά πιο σημαντικό είναι να ελέγξουμε καλύτερα την εφαρμογή των ρυθμίσεων που ήδη υπάρχουν. Πρέπει οι αντιπροσωπείς των γυναικών να έχουν μεγαλύτερο, περισσότερο λόγο στις χώρες αυτές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φροντίσει ακόμα περισσότερο για την ισότητα μεταξύ των γυναικών, την πρόθεση της εκπαίδευσης και άλλα μέτρα. Δηλαδή οι επενδύσεις πρέπει να γίνονται περισσότερο στις γυναίκες για να ενισχυθούν αυτές περισσότερο αλλά και για να μπορέσουν να έχουν το δικαίωμα να γεννηθούν. Θα σας δώσω εδώ τώρα και κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Στην Επιτροπή Γυναικών, που είναι επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή, είχαμε βέβαια συζήτηση και συζητήσαμε για τροπολογία. Σήμερα πρέπει να ψηφίσουν, σήμερα το απόγευμα ψηφίζουν στην Επιτροπή Γυναικών μετά τις 4. Οι τροπολογίες ήταν μέχρι τις 22 Μαΐου, 20 τροπολογίες υποβλήθηκαν και σας ευχαριστώ όλους για τις προτάσεις σας. Τώρα πιστεύω ότι το κείμενο της γνωμοδότησης θα επιφέρει τις αλλαγές που χρειάζονται για να καταργηθεί αυτή η βάρβαρη πρακτική. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και αν θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για τις πρακτικές αυτές, βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας. Μην ξεχνάτε όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν γίνει και ευχαριστώ και την γραμματεία που με βοήθησε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Μίτσελ τώρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κυρία Κρετού για την έκθεσή σας, για την γνωμοδότησή σας αυτή. Σήμερα το πρωί στο BBC λέγαν ότι οι Κινέζοι έσωσαν ένα γοράκι. Αν ήταν κορίτσι, ίσως δεν θα είχε βγει στις ειδήσει με τον ίδιο τρόπο. Και χαίρομαι που βλέπω ότι η συντάκτρια τονίζει ότι ο οι λέει ότι 200 εκατομμύρια γυναίκες λείπουν από τον κόσμο αυτή τη στιγμή εξαιτίας των αυλώσεων που γίνονται ακριβώς επειδή πρόκειται για κορίτσια. Επίσης είναι εκπληκτικό να δούμε πώς έτοιμος είναι ο κόσμος να δίνει συνεντεύξεις και να συζητάει τέτοια πράγματα σαν να είναι απόλυτα φυσιολογικά. Γίνονται εκστρατείε. Ο σεξισμός έχει να κάνει με τα συμφέροντα. Σε χώρες όπως είναι η Ινδία και η Κίνα, όπως είπε και η συντάκτρια πολύ σωστά, τα αγόρια οικονομικά έχουν μεγαλύτερη σημασία, γιατί θα φροντίσουν να κερδίσουν χρήματα για να στηρίξουν την οικογένειά τους. Σε ορισμένες περιοχές της Ασίας δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες για γάμο. Οπότε τώρα βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου αναγκάζονται να απαγάγουν κορίτσια από άλλες περιοχές, να τα μεταφέρουν στις δικές τους για να έχουν ύφε. Οπότε πολύ χαίρομαι που αρχίζουμε να το συζητάμε. Θέλω να σας πω και το εξή. Ας προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για την φιλοκτονία και να το ξεχωρίσουμε αυτό με άλλα θέματα για τα οποία μπορεί να διαφωνούμε. Εδώ νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Μην διαχαστούμε εξαιτία άλλων θεμάτων που συνήθω μας διχάζουν. Ας περιοριστούμε εδώ στη φιλοκτονία αυτή καθεαυτή, στη φιλοκτονία σε βάρος των γυναικών. Ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τους οικονομικούς λόγους που οδηγούν στο φαινόμενο αυτό, στην επιλογή δηλαδή της ε, γέννησης ή όχι ανάλογα με το φύλλο του εμβρίου. Και ας φροντίσουμε να υπάρξει μεγαλύτερη κοινωνική προστασία και να καταργηθεί η προτίμηση αυτή υπέρ των αγοριών. Υπάρχει άμεση σχέση. Υπάρχει το θέμα της ασφάλειας είτε πρόκειται για την υγεία, είτε πρόκειται για τις οδιές. Η πραγματικότητα είναι ότι για ορισμένε από τις οικογένειες που οδηγούνται στις ε, πρακτικές αυτές, η ασφάλειά τους είναι να τον έχουν ένα γόρι. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Και όσο περισσότερα κάνουμε για να αλλάξει αυτό, τόσο το καλύτερο. Και χαίρομαι που βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συζητήσει με ακαδημαϊκούς και μεταφέρουν τις ανησυχίες που έχουν μεταφέρει και διάφοροι εδώ. Ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική ασφάλεια. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, οι οικογένειες αυτές να μην νιώθουν ότι έχουν να χάσουν αν αποκτήσουν κορίτσι αντί για γόρι. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της και ελπίζω ότι όταν θα φτάσει στην Ολομέλεια δεν θα έχουμε τις διαφορές που συνήθως εμφανίζονται εκεί και θα μπορέσουμε όλοι μαζί να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάσμαν. Έχετε το λόγο κύριε Κάσμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Κορίνα Κρετού για την εξαίρετη γνωμοδότησή της, γιατί πραγματικά μπαίνει στην καρδιά του ζητήματος. Όπως είπε και ο Γκέι Μίτσελ, πράγματι είναι ανησυχητικά τα νούμερα. Θα ήθελα όμως, αντί να πηγαίνουμε στο πιο μακριά, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Τι γίνεται. Πετάμε στα σκουπίδια μια ζωή επειδή έχει το λάθος φίλο. Είναι απαράδεκτο. Και προέρχεται από μια νοτροπία που θεωρεί ότι η γυναίκα ανήκει στις οικογένειές της, ανήκει στους άντρες. Αυτό πρέπει να αλλάξει. να αλλάξει νοοτροπία. Εγώ συμφωνώ με τον Γκέ Μίτσελ ότι υπάρχουν λόγοι γνωστοί που υποστηρίζουν μια τέτοια προσέγγιση. Η Κορίν μας υπενθυμίζει τις επιπτώσεις. Οι γυναίκες όμως, αν δεν γεννηθούν, πώς θα αποκτήσουν δικαιώματα, πώς ε, θα γίνουν χρήσιμες στην κοινωνία. Σίγουρα υπάρχει ανάγκη για νομοθεσία. Χρειαζόμαστε νομοθεσία κατά των πρακτικών αυτών επιλογής του φίλου. Και συμφωνώ με τον Γκέι Μίτσελ για το ότι τα διάφορα ζητήματα πρέπει να τα βάλουμε στην πάντα. Εδώ πρέπει ενωμένοι να πάμε κατά της φιλοκτονίας και να μιλήσουμε με μία φωνή στο Κοινοβούλιο προσβλέπω στην ψηφοφορία. Δυστυχώ σήμερα το απόγευμα δεν θα είμαι εδώ, αλλά να ξέρει ότι έχει τη στήριξή μου. Απόλυτα. Χτες το βράδυ, πέρα από τι διάφορες εκθέσει, τι λέει κάτω, λέει ενωμένοι στην διαφορά. Μα αν είμαστε ενωμένοι στη διαφορά, τέλεια. Αλλά από την άλλη μεριά διχαζόμαστε στην ενότητα. Οπότε αυτή τη φορά ας μείνουμε ενωμένοι. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ο Μίκαλ Κούσταυσον, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια, τη συντάκτρια της νομοδότησης για την εξαιρετική γνωμοδότηση. Όπως και οι δύο προλαλήσαντες, πιστεύω και εγώ ότι είναι ανατριχιαστικό παράδειγμα της, ε, του πατριαρχισμού που επικρατεί στη, στην κοινωνία μας. Συνδέεται με το δικαίωμα των ανδρών να ε, λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τα σώματα των γυναικών ε, και αυτό είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει. Και συνδέεται το θέμα αυτό και αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε, συνδέεται με την κοινωνική διάσταση και την δομή της κοινωνίας. Λείπει, για παράδειγμα, ε, η κοινωνική πρόνοια, υπάρχει μεγάλη φτώχεια και γι' αυτό ε, έχει περισσότερο περιθώριο να ε, αναπτυχθεί ο πατριαρχισμός. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν ε, σε όλο τον κόσμο μπορεί να υπάρχει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, αλλά ουσιαστικά υπάρχει παντού. Τα δικαιώματα των γυναικών, το δικαίωμα των γυναικών να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν το σώμα τους, ε, είναι θεμελιώδες δικαίωμα και θα πρέπει να γίνεται σεβαστό σε όλους ε, τους τομείς. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός στο δικαίωμα αυτό. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νιούτον Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, συμμετέχω στην αντιπροσωπεία προς το Ινδικό Κοινοβούλιο. Και είναι συναρπαστικό αυτό, διότι όχι μόνο επισκεφτόμαστε το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο στο Νέο Δελχή, αλλά μαθαίνουμε ότι είναι πολύ αδύναμο το Κεντρικό Κοινοβούλιο και ότι τα 28 κρατήδια της Ινδίας κάνουν ό,τι θέλουν. Ε, ε, είναι αυτό αρκετά παρόμοιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Μια μέρα λοιπόν επισκεφτήκαμε ένα χωριό για να δούμε πώς ε, η επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε σταματήσει τη ε, δουλειά ε, των παιδιών. Ε, και ήταν πολύ συγκινητικό που το είδαμε και ε, συγχαρήκαμε ε, έναν από τους οργανωτές και μας είπε ότι ναι πράγματι τα καταφέραμε αλλά υπάρχουν τόσα άλλα χωριά ε, στην Ινδία όπου δεν έχει γίνει τίποτα. Επίσης επισκεφτήκαμε την Πάτνα που είναι, ε, λέγεται ότι είναι ε, το φτωχότερο κρατήδιο της Ινδίας και στο Δημαρχείο, πράγματι διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ φτωχό το χωριό. Είχαμε λοιπόν στο Δημαρχείο μια συζήτηση που συμπεριέλαβε και το θέμα της ανάπτυξης του πληθυσμού και της και της ε, δολοφονίας των μικρών παιδιών. Ε. Και μας είπαν ότι δεν προσπαθούμε καν να ελέγξουμε ε, την αύξηση του πληθυσμού της Ινδίας, που είναι και αυτό σημαντικό πρόβλημα. Αλλά στη συζήτηση στο Δημαρχείο της Πάτνα. Ε, εγώ καθόμουν να τα, το πίσω μέρος της αίθουσας ε, και ε, δίπλα μου καθόταν μια μορφωμένη Ινδύη κυρία και όταν φτάσαμε στο θέμα της φιλοκτονίας μου είπε... Μου είπε, εγώ ακόμα δεν βρήκα κάποιον άντρα που να, που να είναι διατεθειμένος να το κάνει. Είναι πολύ βαθύ το πρόβλημα λοιπόν στην Ινδία, ε, όπου υπάρχουν αιώνες παράδοσης στην Ινδία. Ε, έχουμε δίκιο λοιπόν που εκπονούμε αυτή την έκθεση, αλλά ε, θα μας πάρει πολύ χρόνο μέχρι να αλλάξουν οι απόψεις, ιδιαίτερα στην υπεθρό της Ινδίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ως σκιώδης εισηγήτρια της ΑΛΔΕ, Μπορώ να συμφωνήσω όσον αφορά ε, την Ινδία ε, και έχει απόλυτο δίκιο ε, για μας τους Ευρωπαίους. Είναι σαφές τι σύστημα αξιών έχουμε και τι θέλουμε να προωθήσουμε στην αναπτυξιακή μας συνεργασία με άλλες χώρες. Το ότι έχουν άλλες χώρες όμως άλλη νοοτροπία είναι άλλο θέμα. Δεν ευχαρίστησα την ε, κυρία Κρετιού για τη γνωμοδότησή της. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, σίγουρα ε, στην περίπτωση αυτή ε, συμφωνούμε και νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε έξω τις ε, κομματικές μας διαφορές γιατί είναι σημαντικό εδώ να προχωρήσουμε ενωμένοι. Στην αναπτυξιακή μας συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να φροντίσουμε να εμποδίσουμε ε, την φιλοκτονία στην ε, Ασία, στην Ινδία, στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Ε, υπάρχει γενική εντύπωση, γενική αίσθηση ότι οι γυναίκες αξίζουν λιγότερο. Εάν ε, ε, αν είχαν καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων, ε, σίγουρα θα ήταν και πιο ισορροπημένη κοινωνία. Ε, αν ε, είχαν μορφωμένε γυναίκε όπω έχουμε εμεί στην Ευρώπη, αν, ε, θα, βλέπανε ότι οι γυναίκε μπορούν να αναλάβουν, να αναλάβουν σημαντικέ θέσει στην κοινωνία. με την εκπαίδευση μπορεί να γίνει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν με την πολιτική να προσπαθήσουμε να ε, του δείξουμε ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Βέβαια αυτό θα διαρκέσει πολύ, έχει δίκιο ο συνάδελφο, αλλά θα πρέπει να επιδιώξουμε ακριβώ αυτό, να πετύχουμε αυτό το στόχο. Έχω υποβάλει τροπολογίε. η μία έχει να κάνει με τους στόχους της χιλιετίας. Η στοχευμένη άμβλωση λοιπόν κοριτσιών είναι σίγουρα κάτι που θέλουμε να καταπολεμήσουμε με τους ε, ε, στόχους της χιλιετίας. Και επίσης όσον αφορά τους, ε, γάμους, ε, τους αναγκαστικούς γάμους ε, παιδιών, και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Ελπίζω λοιπόν ότι θα ψηφίσουμε όλοι ομόφωνα. το θέμα δεν είναι να λέμε ότι απαγορεύεται η αμβλώση. Μιλάμε συγκεκριμένα για τη στοχευμένη άμβλωση κοριτσιών. Ε, θηλυκών εμβρίων. Και θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην υπονομεύσουμε τις εργασίες μας, ε, αλλά να ε, συνεργαστούμε με τους ανθρώπους που επιτόπου φροντίζουν για την εκπαίδευση των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όντω το γεγονό είναι πολύ σημαντικό και έχουμε καθυστερήσει. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μάλλον στην κυρία Γκρέσ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα να στηρίξω την παρέμβαση που μόλις ακούσαμε σε όλες τα σημεία και να υπερθυμίσω την αναγκαιότητα για την υγεία των γυναικών. Αυτό είναι απαραίτητο ως προς την ανάπτυξη και θεωρώ ότι είναι μια μακροχρόνια εργασία, είναι δύσκολη, αλλά είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ε, μακροπρόθεσμες ε, προσπάθειες ε, της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζω τα όσα υπόθηκαν για τον καταναγκαστικό γάμο επίσης σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, γλώσσες κατ' επιλογή. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ το, το δικαίωμα στην άμβλωση θα πρέπει να είναι δικαίωμα για όλες τις γυναίκες στον τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί στο να μην πέσουμε στην παγίδα του να απορρίψουμε κάθε δικαίωμα στην άμβλωση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Κομισιόν, η κυρία Βερτζινή Ραμέλ για δύο λεπτά. Uh, um, πρόεδρε, πρόσφατα την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και συμφωνήσαμε με την Κομισιόν ότι θα καλύψουμε από κοινού το θέμα. Το θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την αξιότιμη βουλευτή για την έκθεση, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και να τονίσω ότι το 2013 είναι μοναδική χρονιά για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε διεθνή φόρουμ και χαίρομαι που ε, ο πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών, κ. Κούσταυσον, είναι παρόν σήμερα στη συνεδρίασή μας. Σε πολλές κοινωνίες όπου το παιδί που γεννιέται μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις ε, στην περαιτέρω ζωή του και να ε, επηρεαστεί με αυτόν τον τρόπο και η ζωή του αλλά και ο θάνατός του, δηλαδή η θανάτωσή του. Να τονίσω επίση ε, πω το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη έχουμε δώσει προτεραιότητα στα θέματα της ισότητας των φύλων. Αυτά μας απασχολούν ιδιαίτερα. Κάνουμε μια προσέγγιση κατάντη ανάντη ε, και τα θέματα της ε, ατζέντα ε, είχαν προταθεί ήδη από το 2009. Τα, οι που αναφέρεται το αξιότιμο μέλος ε νομίζω ότι αναφέρονται ω προτεραιότητε στο πρόγραμμα αυτό. Επίσης αναφίξατε το ζήτημα της συνεργασία με διεθνεί οργανισμού. Εργαζόμαστε πολύ στενά με διάφορε δομέ του ΟΗΕ με οργανώσει των γυναικών έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεννόηση πέρυσι έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει ε, σημαντική ε, απόδοση και στηρίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής σε ζητήματα που αφαιρούνται της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών. Σας ευχαριστώ πολύ, διακόπτη Πρόεδρος. Η Κομισιόν θέλει να λάβει το λόγο. Έχετε δύο λεπτά. Όχι, δεν θέλετε να λάβει το λόγο. Πολύ συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Δώσω το λόγο στην κυρία Κρέτου προκειμένου να συνοψίσει. Ευχαριστώ Προέδρε όπως προείπα. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα για μια ακόμα φορά να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για τις τροπολογίες σας αλλά και για την δουλειά που κάνατε. Αυτό είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα βάρβαρο και έχει σημασία όλοι να έχουμε την αυτή προσέγγιση. Να σας ευχαριστήσω και την Κομισιόν για τα όσα δήλωσε. Πρέπει να έχουμε αυτήν τη διεθνή συνεργασία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί με κάθε χώρα χωριστά όπως είπατε, πρόκειται για θέματα νοοτροπίας. Αυτά δεν είναι εύκολο να τροποποιηθούν με αποφάσεις και ψηφίσματα. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά καθημερινά και ελπίζω να πετύχουμε την επιθυμητή αλλαγή είναι ζήτημα που άφτεται της ζωής εκατομμυρίων γυναικών που έχουν το δικαίωμα να γεννηθούν, να ζήσουν αξιοπρεπώς στον κόσμο μας και να έχουν μια καλή και ωραία ζωή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Υπενθυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα ψηφίσουμε την έκθεση με τις τροπολογίες της φυσικά. Και τώρα περνάμε στο σημείο 13 της μισής διατάξεως. Τη γνωμοδότηση στην έκτη πρωτοβουλία ε, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας ε, των Φίλων πρόκειται για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα. Πρόκειται για ε, μια γνωμοδότηση και ο κύριος Μάικλ Κάσουμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που βλέπω ότι είναι παρόν ο κύριος Κούσταυσον από την Επιτροπή Γυναικών. Ε, χαίρομαι όμως επίσης επειδή συνεργάζομαι μαζί του ε, στην ε, η, ε, ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου για την ισότητα των φύλων. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε το θέμα της φιλοκτονίας με τα βασικά δικαιώματα των γυναικών. Να μην αποφασίζει άλλος τι θα πρέπει να κάνει μια γυναίκα με το σώμα της. Ε, ε, η συζήτηση για ε, τα αναπαραγωγικά, για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι σημαντικό θέμα και σημαντικό είναι και εμείς να γνωμοδοτήσουμε. Ας ξεκινήσω λοιπόν από τη βασική μου θέση ότι ε, τα ε, δικαιώματα που αφορούν σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Αναγνωρίζονται σε πολλέ ε, διεθνεί συμβάσει και πιστεύω ότι εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην στο να αφαιρέσουμε αυτά που μας διαιρούν και να ορίσουμε ε, τα δικαιώματα αυτά και να ε, εγγυηθούμε την, ε, παγκόσμια πρόσβαση σε αυτά. Άντρες, γυναίκες, αγόρια, κορίτσια θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα σώματά τους και τη σεξουαλικότητά τους με τον τρόπο που επιθυμούν. Αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά τη γνώμη μου, είναι βασικά θεμελιώδη δικαιώματα, έχουν να κάνουν με την αναπαραγωγή, το δικαίωμα ε, να ε, ε, παράγεται κανείς ή όχι, έχουν να κάνουν με τη ζωή, έχουν να κάνουν και με το θάνατο. Ε, διότι ε, ε, το να μην αναγνωρίζουν τα δικαιώματα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο των γυναικών κατά τη γέννα και καθώς και σε σεξουαλικά μεταδοτικές ασθένειες για άντρες και γυναίκες. Όλοι θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά χωρίς διακρίσεις και χωρίς να επιβάλλονται οι θέσεις άλλων σε αυτούς. Και το αποτέλεσμα είναι μια πιο παραγωγική κοινωνία και ε, καλύτερες, καλύτερη πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες υγείας ε, και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Όλα αυτά συμβάλλουν στην μείωση της εθνισμότητας των μωρών και των μητέρων τους. Ακούσαμε για τα 200 εκατομμύρια κορίτσια τα οποία δεν γεννιούνται ποτέ. Επίσης πάνω από 250.000 γυναίκες ε, σήμερα πεθαίνουν κατά την εγκυμοσύνη ή τη γέννα κάθε χρόνο. Μία αξιοπιστή μελέτη δείχνει ότι η πρόσβαση σε, στον εθελοντικό οικογενειακό προγραμματισμό μπορεί να μειώσει ε, τις στατιστικές αυτές κατά 20%. Ε, έστω και για κανέναν άλλο λόγο, αυτή είναι μια πολύ καλή στρατηγική δημόσια υγεία. Ε, το να ε, ενημερώνουμε τον κόσμο για τα δικαιώματά τους. Ε, τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνει πρόσβαση ε, στην, ε, στον εθελοντικό, εθελοντικό οικογενειακό προγραμματισμό, εθελοντική πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις, σε εθελοντική πρόσβαση σε αντισυλληπτικά και σε πρόληψη σεξουαλικά μεταδοτικών ασθενειών. Και επίσης, κυρία Πρόεδρε, σημαίνει προσβασιμότητα καθώς ε, και προσαρμογή των υπηρεσιών αυτών στις ανάγκες ε, του ατόμου. Πιστεύω ότι το να δίνουμε προτεραιότητα στις γυναίκες ε, και στους νέους στη διαδικασία αυτή σχετίζεται με την επίτευξη των στόχων μας όσον αφορά την υγεία. Και και δυστυχώς υστερούμε πολύ σε κάποιους από αυτούς τους στόχους ε, και να ε, ε, τονίσουμε και το θέμα που αναφέραμε νωρίτερα, κάποια ε, προτιμητέα κοινωνικά πρότυπα, κάτι που δίνει την δυνατότητα για προγεννητική επιλεκτικότητα ανάμεσα με το φύλλο, κάτι με το οποίο διαφωνώ πάρα πολύ όπως ήδη είπα στον πολιτικό διάλογο και με ε, χώρες εταίρους ε, θα πρέπει να τονίσουμε τα θέματα αυτά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει τις ε, δραστηριότητες των οργανισμών κοινωνίας των πολιτών και εμείς πρέπει να στηρίξουμε το, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι στα προγράμματα αυτά δέχονται επιθέσεις απ' έξω αλλά και από μέσα. Θα πρέπει λοιπόν Δυστυχώς οι δραστηριότητες στον τομέα αυτό συχνά απειλούνται και αμφισβητούνται. Πιστεύω λοιπόν ότι το πολιτικό θεματολόγιο θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται ε, με ε, τους απαραίτητους πόρους ε, και την τεχνογνωσία και αυτός, θα είναι, αυτός είναι συχνά ο μόνος τρόπος να υποστήριζει τα δικαιώματα αυτά στον πληθυσμό κάποιων χωρών. Μια τέτοια ηγετική θέση ε, στην, ε, ε, στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετά το 2015 είναι απολύτως ζωτική σημασίας και στον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο ε, θα πρέπει επίσης να ασχοληθούμε το θέμα στην ε, διάσκεψη κορυφής για τους στόχους μετά το 2015. Τέλος, ε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε, όπως είπε ο κύριος Μίτσελ νωρίτερα, μια επικοδομητική γνωμοδότηση η οποία θα ενσωματωθεί στην έκθεση της Επιτροπής ΦΕΜ. Οι προκλήσεις είναι ίδιες, αλλά νομίζω ότι τελικά οι στόχοι είναι οι ίδιοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μάισινερ, έχετε το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Την τελευταία φορά μακρηγόρησα σχεδόν, ε, ε, αλλά αυτή τη φορά μπορώ να είμαι πολύ σύντομη, διότι συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο Μάικλ Κάσμαν. Πράγματι, ε, η έκθεση αυτή συνδέεται πολύ καλά με την προηγούμενη γνωμοδότηση που είχαμε. Το θέμα εδώ είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ε, και ε, σε εκπαίδευση για τις γυναίκες και για τους άντρες. Και ε, Κυρίω για τους νέους. Ε, αυτό είναι αποφασιστική σημασία ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση ε, στι αναπτυσσόμενες χώρε με τι οποίε συνεργαζόμαστε. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι στηρίζουμε τα θέματα αυτά. Εμένα με εντυπωσίασε το ότι ο Μάικλ Κάσμαν είπε ότι μας συμφέρει όσον αφορά το κόστο και το όφελος η στρατηγική αυτή, διότι όσο, όσο καλύτερη είναι η υγεία του παιδιού και της μητέρας, ήδη από την εγκυμοσύνη, τόσο περισσότερο μπορούμε να ελπίζουμε ε, σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ε, συμφωνώ λοιπόν με όλα όσα είπε ο Μάικλ Κάσμαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκρέσ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Κάσμαν για άλλη μια φορά που υποστηρίζει αυτό το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι μερικές φορές ε, τα νούμερα αξίζουν τόσο όσο και μια καλή ομιλία. 222 εκατομμύρια γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση στην αντισύλληψη. 4,5 εκατομμύρια εγκυμοσύνες ανεπιθύμητες έχουμε κάθε χρόνο και κάθε λίγα λεπτά πεθαίνει μια γυναίκα εξαιτία μια άμβλωση που δεν γίνεται κάτω από ιατρική παρακολούθηση κάθε 11 λεπτά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι πραγματικά πολύ σοβαρό. Έχουμε πάρα πολλές ρυθμίσεις για την υγεία, αλλά είναι όλες πολύ γενικές. Και τελικά καμία δεν λαμβάνει υπόψη την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Γιατί υπάρχει εδώ και το AIDS βέβαια. Γι' αυτό και χαιρετίζω την έκθεση αυτή, η οποία αποτελεί την ευκαιρία να προωθήσουμε το θέμα αυτό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Και πάλι σας ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Ευχαριστώ κύριος Γκούσταυσον. Ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω με τον ε, Κάσμαν και θα τον επενέσω. Είναι δύσκολο να πω οτιδήποτε καλύτερα ε, από αυτόν. Ε, θα είμαι λοιπόν πολύ σύντομος. Ε, συμφωνώ απολύτως με την παρέμβασή του και πιστεύω ότι η πρόταση που έχει υποβάλει είναι εξαιρετική. Χαίρομαι που η Επιτροπή ΔΕΒΕ γνωμοδοτεί στο θέμα αυτό, διότι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το θέμα αυτό συνδέεται με αυτό που συζητήσαμε πριν, συνδέεται με το δικαίωμα των γυναικών να λαμβάνουν να αποφασίζουν ε, για το δικό τους σώμα ε, και να αποφύγουμε τους, ε, τις πατριαρχικές δομές που συχνά αποφασίζουν για τις γυναίκες τι πρέπει να κάνουν με το σώματά τους. Κάτι επίσης καλό στην πρόταση του Μάικλ Κάσμαν είναι ότι συχνά όταν μιλάμε για δικαιώματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία μιλάμε για το δικαίωμα στην άμπλωση. Ε, αλλά τα ε, δικαιώματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι ε, πολύ ευρύτερα από αυτό και το αναφέρει ο Κάσμαν αυτό. Έχει να κάνει με την ενημέρωση, με, τις, ε, με, την αντισύλληψη και λοιπά. Μ' αρέσει λοιπόν η πρόταση του Μάικλ Κάσμαν και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σωστά όλα αυτά που είπε και συμφωνώ απολύτως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πιτσιλίδης έχει τώρα το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ίσως τη γλώσσα μου κι εγώ. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος γιατί ο εξαίρετος συνάδελφος έχει πρώτα απ' όλα κάνει μια πολύ καλή δουλειά και για την οποία θέλω να το συγχαρώ. Και δεύτερο γιατί όλοι οι συνάδελφοι που μίλησαν συμφωνούν και με έχουν καλύψει. Θέλω μόνο να τονίσω κι εγώ από τη μεριά μου ότι μου άρεσε ιδιαίτερα και ξεχωρίζω αυτό που είπε ο κύριος Κάσμαν ότι οι πεπιθήσεις των άλλων δεν μπορούν να επιβάλλονται σε άλλους ανθρώπους. Σε αυτό το σημείο, επειδή στη δική μου πολιτική ομάδα καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί και να αντιδρούν με κάποιες από τις απόψεις που αναφέρονται στην έκθεση αυτή, θέλω να απομακρύνω τις ανησυχίες τους λέγοντας ότι σεβόμαστε είμαι βέβαιος ότι και ο κύριος Χάσμα συμφωνεί, τι πεπιθήσει κάθε ανθρώπου φτάνει να τι επιβάλλει στον εαυτό του και όχι στους άλλους. Αν με αυτό συμφωνούμε τότε νομίζω μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε με αυτή την εξαιρετική έκθεση και να την ψηφίσουμε όλοι μαζί δίνοντας ένα δυνατό μήνυμα προ όλου του λαού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Γκέρντζ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Μία ερώτηση έχω να θέσω. Σκέφτηκε να μας διαφωτίσει σχετικά με τι κάνει το Ταμείο του ΟΗΕ για τον πληθυσμού στον τομέα αυτό, UNFPA, κατά την άποψή μου κάνει μια αξιόλογη εργασία που εκτιμάται από το σύνολο της διεθνούς κοινωνίας, κοινότητας, εκτός από κάποιες περιπτώσεις όπου ε, τυχε επίθεση από πλευρά ΙΠΑ, λανθασμένα φυσικά, διότι κατηγορήθηκε πως διαδίδει και διαχέει των ε, ως μέσο ελέγχου των γεννήσεων στην Κίνα. Αυτό διαπιστώθηκε ότι ήταν κάτι το πριν από μερικά χρόνια αρκετοί από εμά ε, στηρίξαμε τον ρόλο που διαδραματίζει το UNFPA. Δεν έχω σαφείς προφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της δράσης αυτής της οργάνωσης σήμερα, αλλά θα ήθελα να συμφωνήσουμε εδώ στο πλαίσιο Επιτροπής πως πρώτον ο ΙΕ κάνει εξαιρετική εργασία στον τομέα αυτό και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον έχει ικανοποιητικά μέσα. Εδώ μιλάμε για συμπληρωματικότητα στη δράση. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον και η Κομισιόν συμβάλλει στην καλή και χρηστή λειτουργία αυτού του μηχανισμού. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζεύκα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Κομισιόν. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεση και για τις συστάσεις. Όπως ήδη ανέφερα, οι προτάσει σα σχετικά με το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωση είναι σημαντική και ε, πρέπει στη στρατηγική που προωθούμε να λάβουμε υπόψη και το ρόλο τη κοινωνία των πολιτών, που και αυτή παίζει σημαντικό ρόλο, να υπογραμμίσουμε μια σειρά από τους στόχους της χιλιετίας ε, η Υπουργή Ανάπτυξης ε, πρόκειται να συνδυάσουν σήμερα και ένα από τα θέματα θα είναι ακριβώς αυτό το, ζήτημα. Και περιμένουμε οι Υπουργοί να στηρίξουν την πλήρη εφαρμογή της πλατφόρμας του Πεκίνου και το πρόγραμμα δράσης του Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και τα αποτελέσματα των διασκέψεων για το θέμα της αναπαραγωγικής υγείας. Επίσης η Κομισιόν έχει μια πολύ καλή πρόταση για το θέμα της, των, δικαιωμάτων, των αγροτικών δικαιωμάτων. Ίσως να δώσω το λόγο στην, στις υπηρεσίες της Κομισιόν για να μιλήσουν για το πρόγραμμα. Ανέφερε ναι, αρνητικά η Κομισιόν. Να συνοψίζω ότι έχουμε μια σειρά από προγράμματα σε χώρες που στις οποίες αφορά αυτό το πρόγραμμα των δικαιωμάτων για την, στην αναπαραγωγική υγεία. Ευχαριστώ. Η κυρία Τουρίντ έχει δύο λεπτά στο διάθεσή για να μας ενημερώσει σχετικά με το θέμα από την Κομισιόν. Η κυρία Τούρικ δεν είναι παρούσα, θα τα χρησιμοποιήσω εγώ τα λίγα λεπτά. Ευχαριστώ για το έγγραφο. Η Κομισιόν στηρίζει φυσικά την ε, πρόγραμμα δράση του APCD και έχουμε διάφορα προγράμματα που τρέχουν σε επίπεδο κρατών μελών. Ο βασικός στόχος της Κομισιόν είναι να στηρίξει τα συστήματα υγείας των κρατών και να προβλέψει την απαραίτητη ε, παροχή υλικού αλλά και προσωπικού για τους κοινωνικούς τομείς αλλά και για τον τομέα της υγείας. Τώρα σχετικά με το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουμε διάφορα προγράμματα με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε πολλά κράτη την οικοδόμηση ικανοτήτων διαφόρων οργανώσεων για να προβλέψουν την σεξουαλική κατάρτιση και εκπαίδευση, ε, ενημέρωση, συμβουλές ε, και ανακοινώσεις. Ε, επίση. στηρίζουμε το UNFPA. Υπάρχει κάποιο μεγάλο πρόγραμμα το οποίο στηρίζει το συνολικό πρόγραμμα της σεξουαλικής αναπαραγωγικής υγείας Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κάσμαν για μερικά λεπτά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τόσα είπαν και για τη στήριξή τους. Θέλω να απαντήσω σε μερικά πράγματα. Αυτό που υπενθύμισε η κυρία Γκρέις είναι πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα, πόσο τεράστιο είναι ότι οδηγεί σε απώλεια ζώνη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να στηρίξουμε αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διάσκεψη για τα μετά το 2015 είναι μια διάσκεψη στον ΟΗΕ δηλαδή που πρέπει να μιλήσουμε όλοι με μία φωνή. Ο κύριος Γκούστευσον επίσης έχει δίκιο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, νοοτροπίες είτε βασίζονται σε θρησκευτικές απόψεις, είτε πολιτιστικές, είτε οτιδήποτε άλλο. Κύριε Πολιτσίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα είπατε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ακριβώς. Και το λέω ως άθεος. Σέβομαι και τη θρησκεία και όλα. Θεωρώ ότι είναι πολύ ιδιωτικά και προσωπικά. Το πιο προσωπικό και ιδιωτικό δικαίωμα. Αλλά δεν πρέπει ποτέ το δικαίωμα αυτό να το επιβάλλουμε σε κάποιον άλλον. Διότι επιβάλλοντας κάτι μειώνεις το δικαίωμα του ατόμου εφόσον του το επιβάλλεις και δεν μπορεί μόνος του να το αποφασίσει. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε, να αναγνωρίσουμε τις διαφορές και να σεβόμαστε τις πεπιθήσεις και τις ιδέες που έχουν οι άλλοι γιατί παραμένουν του ιδιωτικού και του προσωπικού του τομέα. Ε, ο κύριος Γκέρενς έχει δίκιο όπως πάντα. Τσάρλς, σωστά υπενθυμίζεις την καλή δουλειά που κάνει ο ΙΕ. Όντως γίνονται επιθέσεις, δηλαδή γίνονται προσπάθειες να μειωθεί η χρηματοδότηση από τις Ηνωμένε Πολιτείες και από την άκρα δεξιά το ευαγγελικό που λέω εγώ, την ευαγγελική πολιτική δεξιά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τον ΟΗΕ, να δούμε τι κάνουν εκείνοι, τι ζωές που έχουν ε, σώσει, τι έχουν κάνει για τις γυναίκες, τα αγόρια, τα κορίτσια, όλη τη δουλειά που κάνουν πράγματι. Και ακριβώς επειδή βρίσκονται σε δύσκολη θέση, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να βρεθούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου μαζί τους και να πούν γιατί είναι ζωτική σημασία αυτή η δουλειά. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η Παρασκευή, αν δεν απατώμε. Ίσως όχι. Ευχαριστώ πολύ πάντως το Ρενό το βοηθό μου για το εξαίρετο έργο του όσον αφορά αυτή την υπόθεση. Ξέρετε, όταν κάτι δεν πάει καλά στη δημόσια ζωή τα βάζουμε μαζί τους, αλλιώς τους ξεχνάμε. Πάντως πραγματικά, επειδή με συμβούλεψε τόσο καλά και με βοήθησε τόσο πολύ, έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που έχουμε μπροστά μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η Τετάρτη Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 9 Ιουλίου. Και τώρα είμαστε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο γνωμοδότησης μη νομοθετικού χαρακτήρα που έχει να κάνει με τη διαφθορά στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και τις συνέπειες που έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες. Η συγητής μας, μάλλον συντάκτης γνωμοδότησης, είναι ο κύριος Καμίνσκι, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν μπορεί να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Θα τον αντικαταστήσει ο κύριος Γιάν Σαγραντήλ, στον οποίο δίνω και το λόγο ευθύ αμέσω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ζητήσω να μεταφέρω τι απολογίε του ε, κυρίου Καμίνσκι που δεν μπορεί να είναι παρόν. Θα προσπαθήσω να τον, να τον αντικαταστήσω. Θα προσπαθήσω να είμαι και όσο γίνεται πιο σύντομο, ε, διότι το θέμα αυτό στη, στο σχέδιο γνωμοδότησης ε, δεν είναι τίποτα νέο. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν το πρόβλημα τη Ε, της ε, διαφθοράς στην δημόσια χρηματοδότηση, ιδιαίτερα στον τομέα της ε, αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας ε, που προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά χρήματα ε, χάνονται κάθε χρόνο σε, παράνομα, ε, σε, σε παράνομες χρηματοδοτικές ροές. Σε πολλά χρήματα ε, κρύβονται σε υπεράκτιους λογαριασμούς και έχουμε και άλλες παράνομες συναλλαγές. Όλοι τα γνωρίζουμε αυτά το, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό επανειλημμένο στο παρελθόν. Ε, φαντάζομαι ότι και στο ε, μέλλον θα μας ακόμα. Είναι αρκετά σοβαρό το θέμα αυτό λοιπόν για να επανέλθουμε και να προσπαθήσουμε να ετοιμάσουμε κάτι και να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που να επικεντρώνονται κυρίως ε, στην υποχρέωση λογοδοσίας, την διαφάνεια, στον, όσον αφορά τη χρήση ε, των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που διατίθενται για ε, αναπτυξιακούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Ο κύριος Καμίνσκι έχει υποβάλει μια σειρά προτάσεων. Προτείνει η Επιτροπή Ανάπτυξης να καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της Ε, τις ε, εξής προτάσεις, ε, να τονίσουμε ότι η συστημική διαφορά αποδυναμώνει του κρατικού θεσμού και εξασθενίζει την ικανότητα των κυβερνήσεων να εκπληρώσουν τι υποχρεώσει του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίω σε σχέση με τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των, πολιτικο... των πλέον ευάλωτων και περιθεωριοποιημένων. Επίση, θεωρείται ότι πρέπει να, αναγνωρίζουμε... να αναγνωρίζει η Επιτροπή μα ότι η διαφθορά ε, έχει ω αποτέλεσμα την, κατα... την κακή κατανομή των πόρων ε, και είναι καταστροφική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση τη στόχια, ενώ αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων τη χιλιετία. Ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η διαφθορά είναι παγκόσμιο φαινόμενο και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταπολεμήσει τόσο την εξωτερική όσο και την εσωτερική τη διάσταση, ε, προκειμένου να περιοριστούν οι εξαγωγή εξαγωγής ε, διαφθοράς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης θα πρέπει να σημειώνουμε την ανησυχητική αύξηση του όγκου των κεφαλαίων που διαφεύγουν από τι αναπτυσσόμενε χώρε, όπου τα χρήματα που προέρχονται από τα Ροδοκία θεωρείται ότι ανέρχονται στο 3% περίπου των εκτιμώνων παράνομων χρηματοοικονομικών νερών και να υπενθυμίζουμε ότι μόνο το 2% των παράνομων αυτών ροών επαναπατρίζονται στι χώρε από τι οποίε προέρχονται και επίση να τονίζουμε ότι η πάταξη τη διαφορά εντάσσεται σε ευρύτερε προσπάθειε για την προαγωγή τη χρηστή διακυβέρνηση, η οποία ορίζεται ω μία από τι βασικέ προτεραιότητε για τη βελτίωση τη αποτελεσματικότητα τη αναπτυξιακή βοήθεια Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόγραμμα δράση για αλλαγή του 2011. Και πάλι, Επίσης, ε, να πω ότι η προτάση αυτή του κυρίου Καμίνσκι δεν είναι τίποτα νέο. Το θέμα αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Και ο κύριος Καμίνσκι πιστεύει ότι είναι αρκετά σοβαρό το θέμα ώστε να αναλάβουμε δράση και ως Επιτροπή να προτείνουμε τη λήψη πιο συγκεκριμένων μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι άλλες επιτροπές, ε, ιδιαίτερα η ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, θα πρέπει να ε, συμμετάσχουν. Ζητώ και πάλι συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Καμίνσκι που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί για να παρουσιάσει ο ίδιος την έκθεσή του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Παρακαλώ, κύριος Βάρσεν. Αν θέλετε δηλαδή να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Μετά την έκθεση της Άννας Γκόμες, που παρουσιάστηκε χτες, έχουμε τη δικιά σας γνωμοδότηση τώρα του κ. Καμίσκη και σας ευχαριστώ για αυτήν. Οι πρώτες μου παρατηρήσεις έχουν ως εξή. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε με την κύρια γραμμή που ακολουθεί η γνωμοδότηση αυτή. Όντως, η διαφθορά αποτελεί απειλή και έχει να κάνει με την ακαιρεότητα των κυβερνήσεων και ολοκλήρωσης της κοινωνίας τελικά. Έπειτα, η διαφθορά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να προχωρήσουν στην επικύρωση της σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς. Πιστεύουμε ότι οι μηχανισμοί αναθεώρησης που δημιουργήθηκαν το 2009 ενισχύουν το κοινό μας έργο. Στηρίζουμε επίσης τις ομάδες εργασίας σε διακυβερνητικό επίπεδο κατά της διαφθοράς. Σε επίπεδο τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθαρά. Τη απουσία των συναδέρφων από την DigiHome Home θέλω να υπογραμμίσω ότι έχουμε ένα εύρος δραστηριοτήτων που έχουν μελετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επεξεργάζονται ιδιαίτερα σε σχέση με το πακέτο του 2011 κατά της διαφθοράς. Τέλος. Στην τρίτη παράγραφο της γνωμοδότησης αναφέρεται κάτι για την εξαγωγή της διαφθοράς ε, υπάρχουν ε, πολύ σκληρά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεωρήσει ότι βρίσκεται στην πρώτη σειρά των κρατών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο κύριος Κόρτης Λάστρα έχει λόγο. Ζητώ συγγνώμη Πρόεδρε, λυπάμαι που δεν ήμουν παρόν στην αρχή της συζήτησης, αλλά είχα μια επίσκεψη και βγήκε σε λίγο παραπάνω. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή καταρχάς για την έκθεση και να πω τα εξής. Το έπραξε και η Υπηρεσία Ευρωπαϊκή δράση για την πρόληψη, για την κύρωση αλλά και την εκρίζωση τη διαφθοράς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι μια απειλή την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Επίσης η διαφθορά ξέρουμε πολύ καλά ότι πλήττει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε μορφή του και ιδιαίτερα στι πιο φτωχέ χώρες του πλανήτη σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τα χρήματα που χάνονται είναι 180 φορές περισσότερα από αυτά που θα αρκούσαν για να αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι ικανό εισόδημα. Και όπως καταλαβαίνετε η διαφθορά πλήττει ιδιαίτερα τα παιδιά και τους αφαιρεί τα διατροφή αλλά και το δικαίωμα στη ζωή. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς, να αποφύγουμε διάφορες τρευρώσεις στην οικονομία αλλά και να βελτιώσουμε την ηθική διότι αυτό ε, αυτό πράττει η διαφθορά οδηγεί στην ανηθικότητα. Ως εκ τούτου, η Σύμβαση των κατά της διαφθοράς θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως και άμεσα. Να είμαστε υπεύθυνοι, διάφανοι, αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης συμπεριλαμβάνουν και της εργασία που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ε, ξεκινήσει, έχουμε, μάλλον το μέσο συνεργασίας έχει παραλύσει λόγω των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων που ε, επαιτεί το Συμβούλιο. Τώρα θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία των κυβερνήσεων, των κοινοβουλίων, αλλά και η Κομισιόν θα πρέπει να ξέρει μια κοινή λύση για το πώς θα αντιμετωπιστεί η διαφθορά σε κάθε κράτος μέλος. Να ενισχύσουμε τα κοινοβούλια, την πολιτεία των την κοινωνία των πολιτών και τονίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συνέπεια των πολιτικών ανάπτυξης και άλλες πολιτικές να μην παρεμποδίζουν αυτές τις ανοιξικές πολιτικές. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ισχυρή ε, βούληση για να καταπολεμήσουμε αυτή τη διαφθορά και να ε, τονίσουμε τις θέσεις ε, τις οποίες έχουμε προσυπογράψει τελευταία ως Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του μέσου για την αξιακή βοήθεια και σε ό,τι την την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προκειμένου να καταστήσουμε την κατάσταση βέλτιστη, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να πάρουμε δράσεις αποτελεσματικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο για την καταπολέμηση αυτής της διαφθοράς. Η γενικευμένη διαφθορά ξέρουμε ότι παρεμποδίζει την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάπτυξη σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας μας. η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει μέσω των εξωτερικών δράσεων να αναπτύξει την, ε, την ανάπτυξη καταπολεμώντας ε, της, ε, τη διαφθορά. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Κομισιόν. Είναι δύο πρόσωποι. Ποια από τις δύο θα μιλήσει για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για αυτή την γνωμοδότηση όσον αφορά τις σχέσεις της διαφθοράς με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η γνωμοδότηση καταδεικνύει τα στοιχεία κλειδί και λέει ότι πρέπει να αναλυφθεί η δράση και σε εξωτερικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διαφθορά, εδώ θέλω να τονίσω κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις δραστηριότητες ε, της αναπτυξικής πολιτικής. Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί στοιχείο κλειδί γιατί συνεισφέρει σε πιο δημοκρατική διακυβέρνηση και σε ανάπτυξη, όπως επίσης καταπολεμά και την ένδια. Η διαφθορά είναι πολύ περίπλοκο θέμα, το, είπε, το είπαν αυτό ευρωβουλευτές, αναφέρεται και στη γνωμοδότηση. Η διαφθορά όπως λέει και η γνωμοδότηση, έχει να κάνει με τεράστια ποσά από τις δραστηριότητε διαφθοράς. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, αποσπώνται πόροι οι οποίοι θα μπορούσαν να απευθυνθούν αλλού, για παράδειγμα, να καταπολεμήσουν την ένδια. Όσον αφορά τώρα την πολιτική και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ' αυτού, καταπολεμάμε την ένδια, στηρίζοντας την χρηστή διακυβέρνηση και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Και αυτό φαίνεται και στην ανακοίνωσή μας του 2011, την ατζέντα για την αλλαγή. Και φαίνεται και από τις ανακοινώσεις που έχουμε κάνει σχετικά με τον προπολογισμό. Βέβαια τη διαφθορά δεν πρέπει να την καταπολεμήσουμε μεμονωμένα. Πρέπει να την συνδυάσουμε με τη δημοκρατική διακυβέρνηση. η διαφθορά βασικά είναι η αποτυχία ενός συστήματος όπου δεν υπάρχει ακριβώς χρηστή διακυβέρνηση. Άρα λοιπόν πρέπει να μπορεί να υπάρχει επιβολή του νόμου, εκδημοκρατισμός, καλή διαχείριση των οικονομικών κλπ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι προσεγγίζει τη διαφθορά και σε εξειδικευμένες δράσεις αλλά και γενικότερα όταν πρόκειται για την διακυβέρνηση σε διάφορους τομείς όπου δραστηριοποιείται. Θα μπορούσα να σας δώσω παραδείγματα για το πώς το κάνουμε αυτό συγκεκριμένα, αλλά δεν έχω χρόνο. Οπότε το μόνο που θέλω να κάνω είναι να τονίσω τη σχέση της καταπολέμησης της διαφθοράς σε τρίτες χώρες με τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σαραντήλ για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και πάλι. Ελπίζω ο κύριος Καμίνσκι να μπορέσει να είναι εδώ την επόμενη φορά και να συμμετάσχει στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις για την ακριβή διατύπωση που θα συμπεριληφθεί στη γνωμοδότηση αυτή. Εγώ καταλαβαίνω και είναι πολύ θετικό αυτό ότι κανένας δεν αρνείται ότι είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. και ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα θετικό και καρποφόρο αποτέλεσμα με την γνωμοδότηση αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και ο κύριος Καμίνσκι δίχως άλλο θα συνεχίσει το έργο αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 4η Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 24 Ιουνίου. Και τώρα περνάμε στο σημείο 14. Κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ. Τα θλιβερά γεγονότα της Πέμπτης που μας πέρασαν στον Ήγηρα, επιθέσεις καμικάζι με πολλούς νεκρούς και ομήρους, μας υπενθυμίζουν πόσο μεγάλη σημασία έχει το θέμα αυτό της στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας στην περιοχή αυτής στρατηγικής σημασίας. Μια από τις πιο φτωχές περιοχές του κόσμου. Μια περιοχή που είναι θύμα της ε, κατάρας των πόρων. Γιατί ακριβώς ίσως επειδή έχει τέτοιους ε, πλούσιους πόρους, η χώρα και οι κατοικοί βρίσκονται σε τραγική φτώχεια. Θα συζητήσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Ροατά σε έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχετε το λόγο κύριε Ροάτα για να μας παρουσιάσετε τους κύρους άξονες της γνωμοδότησής σας αυτής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι από το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σαχέλ είναι μια τεράστια υπόθεση, γι' αυτό και έκανε έκθεση πρωτοβουλίας η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και εμείς γνωμοδότηση. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας πω που είμαι περήφανος που είμαι εισηγητής για το θέμα αυτό. Ένα θέμα που είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρον και περίπλοκο. Και σας ευχαριστώ για ό,τι ιδέες μου δώσετε κι εσείς. Το 2013 ήρθε στο προσκήνιο μια περιοχή που γενικά δεν προσέχει ιδιαίτερα η διεθνής κοινότητα. Με την επικαιρότητα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αυτή η περιοχή του Σαχέλ που πάει από τον Ατλαντικό στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι μια περιοχή γεωγραφικά όπου ελοχεύουν πολλοί κίνδυνοι, όπου υπάρχει αστάθεια και πολιτική και ανθρωπιστική. Το Σαχέλ, το είπατε, είναι η πιο φτωχή περιοχή του κόσμου. 18 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από λοιμό, πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά από οξύλιμο. Η παιδική θνησιμότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή, 500.000 περίπου κάθε μέρα χάνουν τη ζωή τους. Παρ' όλα αυτά, οι πόροι υπάρχουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ουράνιο, πόροι οι οποίοι θα μπορούσαν εφόσον εκμεταλλευτούν να δώσουν δυναμισμό και να κάνουν ελκυστική την οικονομία της χώρας. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι. Η κατάσταση είναι θλιβερή. Η πραγματικότητα δεν είναι όμορφη. Υπάρχει εμπορία ανθρώπων σε καθημερινή βάση. Η τρομοκρατία είναι παρούσα κάθε στιγμή. Επιθέσεις, το είπατε και εσείς, είχαμε επίθεση την πέμπτη που μας πέρασε στον Ήγηρα. Οικογένειες από τη Γαλλία είναι όμοιροι. Η τρομοκρατία έχει να κάνει με λαθρεμπόριο ναρκωτικών, όπλων, αλλά και με εμπορία παιδιών. 900 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, μηδέν. 1,2% δηλαδή του ΑΕΠ ε, προέρχεται από τέτοιες δραστηριότητε. Όσον ε, αφορά την ομοιρία, 65 εκατομμύρια ε, δίνει στους τρομοκράτες η δραστηριότητα αυτή. Έχουμε την ΑΚΜΗΝ, την ΠΟΚΑΡΑΜ, τα Σαρντίν, διάφορες οργανώσεις τρομοκρατικές δηλαδή, οι οποίες σπέρνουν τον φόβο και τον τρόμο στην περιοχή και δρούν ανενόχλητες. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για το Σαχέλ, που είναι μια περιοχή πλούσια, αλλά γεωπολιτικά ασταθής χωρίς δικαιώματα. Είναι απαραίτητο να δράσουμε και να αποφασίσουμε συγκεκριμένα μέτρα για το μέλλον. Ήδη ο ΙΕ, με το ΜΙΣΜΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε πιο μακριά να κοιτάξουμε μετά από 20 χρόνια πώς θα είναι η κατάσταση. Αν δεν δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια στην περιοχή, για την ανάπτυξη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε πάμε κατευθείαν στην καταστροφή. Η γνωμοδότησή μου θα κινηθεί γύρω από δύο άξονες. Ο ένας είναι η ασφάλεια και ο άλλος είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν πολλοί εμπορικοί οδοί η έλλειψη ασφάλειας όμως, οι διαμάχες ανάμεσα σε χώρες, σε εθνοτικές ομάδες, σε τρομοκρατικές ομάδες έχουν ε, ε, καταστήσει την χώρα έρμεο της τρομοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρξει όμως ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια. Η προβληματική λοιπόν που έχει να κάνει με την ασφάλεια και την προστασία του κόσμου είναι κάτι αναγκαίο προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι με τις τοπικές αρχές και την κυβέρνηση πρέπει να εκπονήσουμε πολιτικές για να καταπολεμηθεί η εμπορία των ανθρώπων, κυρίως παιδιών, και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Πάνω από 20 εκατομμύρια όπλα κυκλοφορούν στο Σαχέλ. Ενώ αν υπάρχει ασφάλεια θα υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να δείξουμε το παράδειγμα και να προσφέρουμε βιώσιμες λύσεις στον τομέα του ελέγχου και της ασφάλειας, με μια προσέγγιση που να συνδέει την Ευρώπη και το Σαχέλ. Δεύτερος άξονας σας είπα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τις γυναίκες πρώτα απ' όλα. Τα... Να τηρούνται τα δικαιώματά τους. Να μην υπάρχουν οι αναγκαστικοί γάνεμοι. Αλλά να μπορούν να προωθηθούν στη δημόσια ζωή. Έπειτα να κοιτάξουμε τα παιδιά, την προστασία τους, την εκπαίδευσή τους να τα προστατεύουμε από τις απαγωγές που τα οδηγούν να γίνουν ε, στρατιώτες. Ασφάλεια, ε, υποδοχή προσφύγων και γενικά συνθήκες για μια ζωή με υγεία. Ανθρωπιστική πολιτική επίσης χρειάζεται. Εμείς δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αναπτυξιακή πολιτική αν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι μένει πολλής δρόμος ακόμα να κάνουν οι χώρες της περιοχής για να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και την ανασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει, έχει τη στρατηγική της για την ασφάλεια στο Σαχέλ, μια στρατηγική που προτείνει συντονισμένα να δράσουμε για την ασφάλεια και την ανάπτυξη, γιατί είναι γεγονός ότι το ένα δεν μπορεί να πάει χωρίς το άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 2013 όρισε έναν ειδικό εκπρόσωπο για το Σαχέλ, τον κύριο Ντεμαντών και υπάρχει και ομόλογός του Ρωμάνο Πρόντι από τον ΟΙΕ. Είμαι πεπισμένο ότι θα μπορέσουν να προχωρήσουν προς την ανάπτυξη. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, αλλά είναι και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Οπότε οι χώρες είναι πιο ευάλωτες και περιοχή σε εγκληματικές οργανώσεις στο Σαχέλ. Υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα αστάθειας και ανασφάλειας. Πρέπει να δούμε το Σαχέλ σαν μια περιοχή που βρίσκεται κοντά μας και μπορεί να αποτελέσει απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τις επιτρέψουμε να παίξει τον ρόλο που μπορεί εν δυνάμει να παίξει διεθνούς εταίρου. Για αυτούς τους λόγους η δουλειά μας πρέπει να είναι φιλόδοξη, συγκεκριμένη, σύγχρονη, να καλύψει ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων και κυρίως να λέει την αλήθεια. Πρόεδρε, για το Σαχέλ έχουμε μεγάλες πολιτικές ε, φιλοδοξίες προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα για πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή. Είμαι πεπισμένος ότι θα δώσουμε μια ισορροπημένη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ζωντανή, με απαντήσεις για όλες τις προκλήσεις. Περιμένω από εσά, αγαπητοί συνάδελφοι, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας που θα λάβω υπόψη μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γκέρνς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ να συγχαρώ τον εισηγητή που έκανε μια παρουσίαση εξαιρετική τονίζοντας ε, τα σημαντικά ζητήματα και ιδίω το ζήτημα της ασφάλειας και της ανασφάλειας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να αναφερθώ σε τρία-τέσσερα σημεία. Υπάρχει μια σταθερή σχέση ανάμεσα στην φτώχεια και την ασφάλεια. Δεν πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, όλοι το γνωρίζουμε. Τώρα, σε αυτόν τον φαύλο κύκλο έχουμε όχι μόνο μια κρίση κράτους, αλλά καμιά δεκαπενταριά κρίσεις παρόμοιας φύσης, διότι πολλά κράτη δεν μπορούν να αναλάβουν και να εφαρμόσουν τα δικαιώματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διασφαλίσουν την ασφάλεια και αυτό χρειάζεται μια σειρά από προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρωθούν εκ των προτέρων. Δεύτερον, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κρίση σε επίπεδο περιφερειακής συνεργασίας. Εδώ να τονίσω τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευθύνη της. Η Κομισιόν στην ατζέντα της ε, για το μέλλον έχει τονίσει στην ε, εστίαση της Κομισιόν σε τρεις τομείς και θεωρώ πως αν υπάρχει ένας τομέας ο οποίος ε, ε, αφορά τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η περιφερική συνεργασία που είναι ουσιώδης η ε, Ευρωπαϊκή Συνεργασία, που είναι ουσιώδη σημασία, διότι τα προβλήματα αυτά δεν άπτονται μια χώρα, αλλά αφορούν στο σύνολο τη περιοχή. Πάντω, απέναντι σε αυτή την παρατήρηση που είναι θλιβερή και απογοητευτική, θα ήθελα να αναφέρω και κάποια πλέον ή δράσεις που καλούμεθα να αναλάβουμε, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, εγγράφονται σε ό,τι φορά το άμεσο παρελθόν στο διεθνές δίκαιο. Μόνο η Γαλλία αντέδρασε με τρόπο έντιμο στην πρόκληση που είχε προκύψει πριν από ένα χρόνο για την κατάσταση που επικράτησε στο Μαλί. Θα πρέπει να ε, φόρο τιμή στην Γαλλία και θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς παρόμοιες δράσεις διότι όταν βλέπουμε κάποια δικαιώματα του ανθρώπου τα οποία παραβιάστηκαν στο Μαλί ιδιαίτερα στην νότιο περιοχή του Μαλή. Δεν μπορώ να βρω επίθετο για να περιγράψω αυτή την κατάσταση, δεν λοιπόν, μπορώ να την χαρακτηρίσω. Ε, δεύτερον, η διαφοροποίηση που αφορά στην μελλοντική ατζέντα για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τονίσει περαιτέρω τις προτεραιότητές μας σε ζητήματα σχέσεων με τις χώρες της περιοχής. Εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Υπάρχουν έλλειψη μέσων και η βάση πάνω στην οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί να αναπτυχθούν τα κράτη-μέλη χαρακτηρίζονται από μια πολύ υψηλή γεννητικότητα. Δεν είδαμε ποτέ στο παρελθόν τέτοιο υψηλό ποσοστό γεννητικότητα. Αν έχετε λοιπόν 3% ανάπτυξη, η ανάπτυξη είναι μηδενική, διότι ε, καλύπτεται από την ε, δημογραφική ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά όμως η περιοχή αυτή έχει τεράστιους ε, πόρους. Εδώ σε εκ τούτου υπάρχει ένα έργο, ένα καθήκον το οποίο χρειάζεται να τύχει ιδιαίτερη προσοχή. Ξέρω ότι η υπηρεσία εξωτερική δράση το γνωρίζει. Είμαστε κατάλληλοι για να ενεργήσουμε περί αυτού. Θα πρέπει λοιπόν υπό το φως των αρχών που περιέχονται την ατζέντα της ε, χιλιετίας να εκτιμηθούν αποτελεσματικότερα και καλύτερα διότι αφορά, αφορούν και τη δική μας ασφάλεια, τα δική μας συμφέροντα με την ευγενή έννοια του όρου. Ευχαριστώ κύριε Λέβη, είναι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω και να, συγχαρώ, και να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική παρουσίασή του. Πιστεύω ότι αναφέρθηκαν πολλά θέματα και ο κύριος Γκέρενς τόνισε την σχέση ανάμεσα στη φτώχεια και την ασφάλεια. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί εδώ. Θα μπορούσαμε επίσης να τονίσουμε περισσότερο τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιφέρεια αυτή. Και σκέφτομαι δύο συγκεκριμένα σημεία όπου έχουμε άμεσες επιπτώσεις στην ευημερία και την ε, ασφάλεια παροχής ε, τροφίμων. Η μία περίπτωση είναι η Συμφωνία Αλίας με τη Μαυριτανία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε θετικοί απέναντι στην ανάπτυξη των ε, συμφωνιών αλληλείας, διότι για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διαπραγματεύτηκε συμφωνία αλλιές με τη Μαυριτανία, όπου σέβεται τις ανάγκες των τοπικών αλλιέων και τα δικαιώματά τους για την αλλία οχταποδιών. Αυτό έχει αμφισβητηθεί στο Κοινοβούλιο. Θα ε, ψηφίσουμε αύριο στην Επιτροπή Αλίας ε, για το θέμα αυτό και πολλοί ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι το νέο αυτό πρωτόκολλο δεν περιλαμβάνει ε, ευκαιρίες αλίες για το χταπόδι. Αλλά εάν θέλουμε να στηρίξουμε την ε, βιώσιμη ανάπτυξη σε κάποια μέρη του κόσμου θα πρέπει να σεβαστούμε τις επιθυμίες αυτών των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών. Έχω επισκεφθεί τη Μαυριτανία. Πραγματικά γνωρίζω ότι το θέλουν αυτό και έχω δει και την που δημιουργούν η Αλκάιδα και η Αλσαμπάπ. Είναι πολύ παρούσα η Αλκάιτα και αν θέλουμε να έχουμε σταθερές σχέσεις με τις χώρες αυτές, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να διατηρούμε απεικιοκρατική στάση και να λέμε ότι θέλουμε πρόσβαση στα ψάρια σας. Νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αλλά πιστεύω ότι η ε, έκθεση αυτή περιλαμβάνει και τη Δυτική Σαχάρα στο πεδίο εφαρμογής της. Όχι. Μάλιστα, κρίμα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έλαβα εγώ από συνάδελφο στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Αλλά να αναφέρω, μια και είμαστε εδώ, ότι Μινούσο που ακόμα παρακολουθεί το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας από το 1991 και μετά, είναι η μόνη αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει εντολή που να και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για την σταθερότητα της περιφέρειας αυτής, ότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας μετά από τόσο χρονικό διάστημα. είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πολύ ε, την όλη υπόθεση. Το ότι το θέμα αυτό δεν έχει λυθεί και αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι η Συμφωνία ΛΥΑΣ έχει ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά το Μαρόκο δεν το έχει δεχτεί αυτό όσον αφορά τη Δυτική Σαχάρα. Αυτή ήταν οι παρατηρήσει μου. Ευχαριστώ. Thank you very much for underlining once more the... Ευχαριστώ. Ναι, Όντω η συνοχή έχει τεράστια σημασία όταν πρόκειται για τις διάφορες εξωτερικές μας πολιτικές. Καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε. Τώρα, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ο κύριος Ζερόμ Σπινόζα. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου με τις χώρες της περιοχής. Θα είδατε τα συμπεράσματα του χθεσινού Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η συμφωνία για την προστασία των πληθυσμών και τον σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων. Τονίσαμε σε αυτά τα συμπεράσματα την σημασία της καταπολέμησης ε, της ατιμορρησίας και την άσκηση του κράτους δικαίου στις χώρες της ε, περιοχής. Εξάλλου υπήρξε και ανταλλαγή απόψεων ε, στις 16 Μαΐου με τον πρόεδρο Τραωρέ που ήρθε εδώ ενώπιον σας και μίλησε για το συγκεκριμένο ζήτημα <clears throat> σχετικά με το Μαλί ε, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, ιδιαίτερα στον διάλογο που διεξάγουμε με την χώρα αυτή, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά καθεαυτά, αλλά και τα υπόλοιπα δικαιώματα, αλλά και σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που ο μη σεβασμός του θα μπορούσε να έχει για τις γειτονικές χώρες και η επέκταση της ε, διένεξης στα γειτονικά κράτη Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου αλλά και στο πλαίσιο του μέσου εξωτερικής συνεργασίας. Γνωρίζετε πως υπάρχουν μια σειρά από ε, που προωθούνται. Είμαι σίγουρος ότι η Κομισιόν θα πει περισσότερα πράγματα περί αυτών που αφορούν τόσο μια επιτήρηση από πλευράς αφρικανικής ε, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και σε θέματα δικαιοσύνης, ε, ανθρωπιστικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένου και του μέσου σταθερότητας για την προαγωγή της ειρήνης και της συμφιλίωσης. Η Γενική Προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως προς το Σαχίλ προωθείται σε όλες αυτές τις πτυχές και αυτό υπόθηκε ήδη και από τον κύριο Σιγητή διαπέτε από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ανάπτυξη του Σαχέλ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο Ζερόμ που θα σας μιλήσει λεπτομερέστερα για αυτή τη στρατηγική. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Κάρλ εργάζομαι μαζί με τον συντονιστή για το, για το Σαχέλ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπε ο Κάρλ κάτι ότι δηλαδή δουλέψαμε για την ανθρωπιστική κατεπίκουσα κατάσταση στην Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και ασχοληθήκαμε με τους ε, εσωτερικά ε, εκτοπισμένους ε, αλλά και με τους πρόσφυγες ε, τα τελευταία δύο χρόνια. Οι προσπάθειες έχουν καταβληθεί και αφορούν φυσικά τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών αυτής της περιοχής, το δικαίωμα στην επιβίωση με λίγα λόγια. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα τα θέσανε στο επίκεντρο μια σειράς δράσεων σε θέματα ασφαλείας. Νομίζω πως ο κύριος καθηγητή μίλησε για την ανάπτυξη της στρατηγική UTM. Ε, οι ένοπλες σειράξει αντιμετωπίστηκαν ε, με τρόπο αποτελεσματικά κάτοικοι του Μαλή κατάλαβαν ε, άμεσα την ανάγκη είχαν ε, πολλά να κερδούσουν και αυτό το έκαναν άμεσα κατανοητό. Το το δικαίου που ε, αφορά με θεμελιώδη αντιμετώπιση της δημοκρατίας έχουμε μια δικαστική προσέγγιση στην Ευρώπη διαφορετική το το κόστος των δικαιωμάτων τι είναι να ζητάει από τα κράτη, από το, τα της Σαχέλ να εξαγάγουν έρευνες, συλλογή ε, ευρημάτων και προφοριών σύμφωνα με την τήρηση των κανόνων προκειμένου οι να είναι δίκαιοι και τελικά η πολιτική αποτελεσματικότητα αυτού τους ε, κατά πολέμηση της τρομοκρατία να αποδώσει. Και τώρα κάτι ακόμα για την ε, προσέγγιση, την μακροπρόθεσμη στρατηγική του Σαχέλ που δεν θα ήθελα να φέρω στου τέσσερι πυλώνε εδώ, δεν ξέρω αν υπάρχει λόγο να το πράξω, στοχεύει σε μια δράση που εγγράφεται τουλάχιστον για την προσοχή δεκαετία ή εικοσαετία. Ε, γνωρίζουμε την δημοκρατική έκρηξη και τους λόγους που άπτονται αυτής. Υπάρχουν χώρες ε, που συνορεύουν, η Μαυριτανία, το Μαγκρέμπ, δεν θα χρειάζεται να πείσω τον εισηγητή. Νομίζω ότι γνωρίζουν πολύ καλά την γεωγραφία στην περιοχή η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι να ενταχθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Υπάρχει δυσκολία να αντιμετωπιστεί το θέμα. Η ε, ε, δεν καλύπτει το Μαγκρέμπ, το Μαγκρέμπ δεν παρέχει βιώσιμες δομές και αυτή είναι μια από που ο ειδικό απεσταλμένος έχει εντοπίσει προκειμένου να δουλέψει μακροπρόθεσμα πάνω στο θέμα. Υπάρχει επίσης και το ζήτημα της Λιβύης που είναι κάτι πιο βραχυπρόθεσμο, αλλά συνδέεται με όλες αυτές τις δυσκολίες, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον, αυτόν τον νέο θύλακα ε, αστάθειας. Υπάρχει το ζήτημα των πολυσάριων που κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Γουάντα για να κλείσουμε το θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Δεν θα απαντήσω σε όλους, αλλά μπορώ να σας πω ότι ήδη την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή σήμερα είναι η αρχή, θα έχετε το σύνολο του φακέλου. Θα λάβω υπόψη φυσικά όλες τις παρατηρήσεις που ακούσαμε και θα σας διαβιβάσω νομίζω την 26η ε, την 25η Ιουνίου όλες τις τροπολογίες, ε, η διορθηνη προθεσμία. Πιστεύω ότι ο φάκελος αυτός είναι τόσο σημαντικός και θα ήθελα, όπως είπε ο κ. Κάσμα σήμερα το πρωί, να μπορέσουμε να μιλήσουμε με μία και μόνη φωνή ως Ευρώπη. Αυτό θα αυξήσει την αξιοπιστία μας σε αυτή την ταραγμένη περιοχή. Απαντήσω στο ερώτημα σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα. Επιτρέψτε μου δύο δευτερόλεπτα. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Αυτό το ζήτημα Έχουμε οροδότηση για το Μαλί, την Πουλινοφάσιο, το Τσάντ και όλες τις άλλες περιοχές δηλαδή, που αφορούν την Νότια Σαχάρα. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ε, και νομίζω ότι η Κομισιόν το έθεσε το ζήτημα. Θα πρέπει μια και καλή να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα τάφη. Μίλησα για το Μαρόκο, θα μπορούσα να μιλήσω για την Αλγερία, για την Τινησία. Αποτελούν ένα σύνολο. Εμείς ε, ίσως ε, να κάνουμε μια παράλληλη εργασία, αλλά το παράλληλα δεν συναντώνται ποτέ, δεν συγκλίνουν. Ε, και δεν μπορούμε να αυτοκανικανοποιηθούμε με κάτι το οποίο κάνουμε σε μια περιοχή, αλλά πρόκειται για ένα σύνολο περιοχής. Πάνω από 25 χρόνια ασχολούμαι με το ζήτημα αυτό και το γνωρίζω πολύ καλά από συναδέλφους ε, ότι είμαι στη διάθεσή τους και επιθυμώ, όπως είπα και πιο λίγο, ότι ε, ήμουν υπερήφανο που μου αναθέσατε αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να δώσουμε την εντύπωση ότι η Ευρώπη δίνει ε, ε, την ίδια και τη μεγάλη σημασία στον φάκελο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι θα ακουστείτε και θα υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 25 Ιουνίου στις 6 και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο που είναι το σημείο 16 στην ημερήσια διάταξη. Τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και της οδηγίας της Ευρωπαϊκής σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ένα νομοθετικό θέμα αυτό, πολύ σημαντικό για τις υποανάπτυξη χώρες. Πρόκειται για τα βιοκαύσιμα, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την χρήση γης και την πρόσβαση στη γη. Αγροκαύσιμα θα έπρεπε να το, νομίζουμε, θα έπρεπε να το ονομάζουμε γιατί με την χρήση της γης πετυχαίνουμε τα κάψιμα αυτά. Πριν από ένα μήνα, ο ειδικό εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στην τροφή, ο κύριος Ντεσχιούτερ, εξέφρασε με σημείωμά του τη 23 η Απριλίου για τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή πρακτική των ε, βιοκαυσίμων και ε, για το δικαίωμα στην διατροφή. Εξέφρασε λοιπόν την βαθιά του ανησυχία σε σχέση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκαύσιμα. Μα ζητάει να περιορίσουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους στον τομέα αυτό και να τους εγκαταλείψουμε μάλιστα. Ο κύριος Κασμάρεκ είναι ο εισηγητής μας συντάκτης της γνωμοδότησης, δηλαδή που ετοιμάζουμε για την Επιτροπή Περιβάλλοντος που είναι και αρμόδια επί της ουσίας. Κύριε Κασμαρέκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, συμφωνώ και εγώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το θέμα. Κατάλαβα και εγώ ότι τα συμφέροντα τα οποία διακυδεύονται εδώ είναι πολύ σημαντικά. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, ο τομέα ολόκληρο, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην γνωμοδότηση και στην έκθεση αυτή, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει πόσο μεγάλη σημασία έχει το θέμα. Τώρα, η δικιά μου η άποψη είναι η άποψη και της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης. Αυτήν βέβαια εκπροσωπώ στην γνωμοδότηση. Πρέπει να θυμηθούμε τον αρχικό στόχο της οδηγίας αυτής και τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να τροποποιηθεί η αρχική οδηγία. Αρχικός στόχος λοιπόν δεν ήταν να προωθήσουμε ούτε να αυξήσουμε τα βιοκαύσιμα στην ενεργειακή παλέτα. Ο αρχικός στόχος ήταν να περιορίσουμε τις ε, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τα βιοκαύσιμα λοιπόν δεν αποτελούν αυτό σκοπό, είναι ένα εργαλείο που θέλουμε να έχουμε στη διάθεσή μας για να πετύχουμε τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και γενικότερα αερίου του θερμοκηπίου. Πολύ σημαντικό αυτό γιατί έτσι βλέπουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητάμε για τα βιοκαύσιμα τα οποία περιορίζουν πράγματι τα αέρια του θερμοκηπίου. αλλά λιγότερο από ό,τι είχαμε ελπίσει στην αρχή. Ο ρόλος τους δηλαδή, δεδομένου του στόχου μας του αρχικού, είναι περιορισμένος. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι αποψηλώνουμε για να πετύχουμε βιομάσα ή χρησιμοποιούμε γη η οποία θα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τροφίμων. Και άρα παίρνουμε εδάφη για τα βιοκαύσιμα. Η αλλαγή τώρα στη χρήση γη δεν λάβει υπόψη της ότι βιοκαύσιμα καλλιεργούνται στα εδάφη αυτά. Όταν υπολογίζουμε δηλαδή τις ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου, η βιομάσα που γίνεται καύσιμο όταν ξετάσουμε αυτό το φαινόμενο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις εκπομπές που οφείλονται στην μεταφορά της βιομάζας αυτής. Και αυτό θα έπρεπε να το λάβουμε υπόψη μας. Άρα το όλο θέμα πρέπει να μας προβληματίσει διαφορετικά. Τα βιοκαύσιμα σέβονται τελικά λιγότερο το περιβάλλον και προστατεύουν λιγότερο το περιβάλλον από ό,τι είχαμε φανταστεί αρχικά. Διαπιστώνουμε ότι ο αρχικός μας στόχος συνεπώς δεν επιτυχάνεται μέσω της παραγωγής βιοκαυσίμων και καλλιέργειες όπως είναι το σιτάρι ή ο αραβόσιτος διαθέτουν τελικά λιγότερες εκτάσεις. Οπότε είμαστε στο δίλημα τι να προτιμήσουμε, τρόφιμα ή καύσιμα. Σχεδόν όλη η βιομάζα την ε, παίρνουμε από εδάφη τα οποία χρησιμοποιόντουσαν πριν για τρόφιμα. Άρα υπάρχει ένα ανταγωνισμό εδώ πέρα ανάμεσα στην παραγωγή βιοκαυσίμων και την παραγωγή τροφίμων. Η παραγωγή βιομάζας για βιοκαύσιμα απαιτεί συχνά αλλαγές οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τους παραγωγούς, οι οποίοι είναι συνήθως μικροί παραγωγοί... που δεν έχουν καν τίτλους ιδιοκτησίας των γιών που χρησιμοποιούν, των λιβαδιών που χρησιμοποιούν για ε, τις καλλιεργίες τους, τις αγροτικές τους δραστηριότητες. Έπειτα υπάρχουν τρίτες χώρες, οι οποίες καταλήγουν σε συμφωνίες μεταξύ τους, αλλά τελικά οι αρχικοί χρήστες της γης δεν μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και να χρησιμοποιούν τη γη. Εδώ λοιπόν έχουμε επιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη, αρνητικά επηρεάζουν την ανάπτυξη. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε προοπτική και ναι μεν να αναπτύξουμε περισσότερο την παραγωγή βιοκαυσίμων, αλλά όχι σε βάρος τη παραγωγής τροφίμων. Έπειτα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι οι αρχική αυτοί παραγωγή πρέπει να επιβιώσουν, ενώ τώρα δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη γη και να προωθήσουμε μία προσέγγιση υπέρ των βιοκαυσίμων που να μειώνει πράγματι τις εκπομπές αεριότητα θερμοκηπίου. Αν τα πετύχουμε αυτά, τότε το περιβάλλον δεν θα υποφέρει από την παρετέρω ανάπτυξη των βιοκαυσίμων. Αυτό λοιπόν θα ήθελα εγώ να τονίσω και αυτά προσπαθώ να πετύχω μέσα των τροπολογιών μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τάιλερ έχει τώρα το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε ε, Κασμολέκ. Μιλώντας στην Επιτροπή Ανάπτυξης ε, για τα βιοκαύσιμα, νομίζω ότι ε, πιο σωστό είναι να επικεντρωθούμε στο ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων ε, έχει συνέπειες στις αναπτυσσόμενες χώρες και την πρόσβασή τους σε τρόφιμα. Μιλάμε για 9 δις ανθρώπων μέχρι το 2050 και οι άνθρωποι των υποσυτισμένων ε, αυτή τη στιγμή ε, ανέρχεται σε 873 εκατομμύρια. Πιστεύω λοιπόν ότι η γη θα πρέπει να χρησιμοποιείται για παραγωγή τροφίμων ε, και όχι για να μπορούν οι πιο πλούσιες αναπτυγμένες χώρες να μπορούν να χρησιμοποιούν τα καύσιμα αυτά για τα αυτοκίνητά τους. Λαμβάνοντας υπόψη μου την προσέγγιση του κυρίου Κασμάρεκ ε, όσον αφορά την οδηγία. Ε, αναζήτησα συμβουλές και πληροφορίες ε, και μία από τις πιο σκόπιμες παρατηρήσεις ήταν το Ολιβία που είναι ο ειδικό εισηγητής για το δικαίωμα τροφίμων στα Ηνωμένα Έθνη. Πέντε θέματα βασικής ανησυχίας αναφέρει που σχετίζονται ιδιαίτερα με την συζήτησή μας σήμερα που έχει να κάνει με τα βιοκαύσιμα την, ε, ε, την, ε, την επιρροή τους όσον αφορά την εκρίζωση εδαφών, την ασφάλεια τροφίμων, την έμεση αλλαγή χρήση της γης και την αλλαγή του κλίματος. Κάθε ένα από τα θέματα αυτά θα σας εξηγήσω, γιατί θα προσπαθήσω να τα καλύψω με τις τροπολογίες μου. Ο κύριος Δεσούτα λέει για τα βιοκαύσιμα και την και την εκρίζωση καλοαργαίων. Η ε, καλλιέργεια βιοκαυσίμων ε, απαιτεί μεγάλες εκτάσεις, δημιουργεί κίνητρα ε, για την εκμίσθωση γεών, ιδιαίτερα στην υποσαχαρία Αφρική, όπου δεν προστατεύονται τα δικαιώματα χρήσης της γης. Η τροπολογία υπαριθμών 5, η δική μου, εξηγεί ότι τα βιοκαύσιμα ε, έχουν λάβει περίπου 10 ε, δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο ε, σε δημόσιο χρήμα και γι' αυτό το σύνολο της παραγωγής βιοκαυσίμων το 2020 θα προέρχεται από καλλιέργειες σε γη που, σε εκτάσεις που θα μπορούσαν να, ικανοποιήσουν, να καλύψουν τις αγορές τροφίμων και ζωοτροφών θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε αυτό υπόψη μας ε, όσον αφορά δηλαδή την έμεση αλλαγή χρήση της γης. Ε, υπονομεύεται έτσι η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις εκπομπές. Για να αποφύγουμε λοιπόν την αρπαγή της γης θα πρέπει να γίνει η διάκριση ανάμεσα στις ελαιούχες καλλιέργειες, ε, τα δημητριακά, ε, τα, ε, τη ζάχαρη και άλλες καλλιέργειες για ενέργεια. Η δεύτερη ανησυχία του είναι η ασφάλεια παροχής των τροφίμων. Με, την, με τον καθορισμό δεσμευτικών στόχων ε, και με την επιχορήγηση των βιοκαυσίμων ε, ουσιαστικά ε, οδηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κερδοσκοπία εις βάρος της καλλιεργήσιμης γης. Ιδιαίτερα κοντά σε πόλεις και αεροδρόμια και η αύξηση των τιμών της γης απειλεί τους μικρούς καλλιεργητές σε κάτι που έχει πιθανότατα και αρνητικέ ε, συνέπειες ε, στην ε, ασφάλεια παροχή τροφίμων στι τοπικέ κοινωνίε. Επίση, έχουν έχει αυξηθεί η, η μη σταθερότητα των τιμών των τροφίμων λόγω της αύξησης κινήτρων καλλιέργειας βιοκαυσίμων. Ο κίνδυνος λοιπόν Το θέμα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο δεσμευτικός στόχο ε, του 10% της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκαύσιμα. Επίσης, στην τροπολογία μου υπάρχει μόνο 9 για να μειώσουμε, για να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές ε, συνέπειες ε, όσον αφορά την κερδοσκοπία της γης, για να, χωρίς να περιορίσουμε τη γενική χρήση των βιοκαυσίμων να μπορούν να συνυπολογιστούν ε, Ο συνυπολογισμός ε, για ε, τον στόχο της οδηγίας 2009 κάθετος 28 να μειωθεί βαθμία μέχρι το 2020 όπου θα μηδενιστεί. Και το άλλο θέμα είναι η εκρίζωση της στόχιας και ο κύριος Τεσούτα εξήγησε ότι οι πολιτικές βιοκαυσίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευνοούν ε, τα μεγάλα βιομηχανικά πρότυπα, βιομηχανικής κλίμακας πρότυπα ε, στην Γεωργία. Ε, χρειάζεται δηλαδή περισσότερο κεφάλαιο για τις καλλιέργειες βιοκαυσίμων, κάτι λοιπόν που έχει περιορισμένα ωφέλη για τους τοπικούς πληθυσμούς του Ναντίον. Είναι κάτι το οποίο ευνοεί τους μεγάλους διεθνείς επενδυτές. Ε, αυτό ουσιαστικά λοιπόν ε, ε, είναι αντίθετο με το επιχείρημα ότι τα βιοκαύσιμα θα επιφέρουν επιπλέον κέρδος για τους μικρούς παραγωγούς. Έχω μια συγκεκριμένη τροπολογία η οποία αφορά την καρδιά του θέματος. Ο Διεθνής Οργανισμός ε, Τροφίμων ε, και Γεωργίας αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της ε, δεν είναι βέβαιο ότι θα ευνοήσει τους στοχούς των αντίον. Η γεωργική ανάπτυξη θα πρέπει να ωφελήσει τους μικρούς παραγωγούς. Λένε λοιπόν ότι οι επενδύσεις στη γεωργία είναι τρεις φορές πιο αποτελεσματική από άλλες ε, επενδύσεις για τη μείωση της φτώχειας. Γι' αυτό πολύ σωστά είπαμε ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων υπονομεύει την εκρίζωση της φτώχειας. Όσον αφορά την έμεση αλλαγή χρήσης της γης, ε, το λεγόμενο ILUC, ε, έχω την ε, τροπολογία μου υπαριθμών 12, ε, όπου τονίζω τη σημασία η έμεση αλλαγή χρήσης της γης να... Μάλλον όταν λαμβάνονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου να λαμβάνονται και οι εκπομπές που προκαλούνται από την αλλαγή χρήσης της γης. Και τέλος, όσον αφορά την ε, αλλαγή του κλίματος, ο κύριος Δεσούτα λέει ότι η υπόθεση ότι η πολιτική βιοκαυσίμως Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί σε μείωση ε, των εκπομπών ε, είναι αμφίβολη. Εγώ θα το έλεγα πιο σκληρά. Ιδιαίτερα τα βιοκαύσιμα από σόγια, ελαιοκράμβη και ε, φίνικες ε, ουσιαστικά ε, οδηγεί σε περισσότερες εκπομπές. Αντί λοιπόν να βελτιώνουμε τα πράγματα, τα κάνουμε χειρότερα. Αυτές λοιπόν οι ανησυχίες μου επίσης αποτελούν τη βάση για τις άλλες μου τροπολογίες και προσλέπω στην καλή συζήτηση μαζί σας σε αυτό το χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τόγια έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ευγένεια που επικρατεί στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω με την ευκαιρία αυτή πως η αναθεώρηση των δύο οδηγιών είναι πολύ σημαντική και μας δίνει ιδιαίτερη ευθύνη ως Επιτροπή διότι η εξέταση που θα κάνουμε ε, αφορά έναν κλάδο ο οποίος δεν έχει τύχει σαπέρα της προσοχής ε, για αυτή την πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ευστήσουμε την προσοχή όλων των άλλων ε, επιτροπών σχετικά με την ανάγκη συνοχής, και συνέπεια που θα πρέπει να υπάρξει με τις πολιτικές μας, δηλαδή συνέπεια και συνοχή με τις ενεργειακές πολιτικές, πολιτικές περιβάλλοντος που είναι ιδιαίτερα σημαντική ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική ε, την αναπτυξιακή και η αναθεώρηση των άλλων προσεγγίσεων, άλλων οδηγιών βλέπετε από άλλη οπτική γωνία. Και εμείς λοιπόν θα πρέπει να συντονίσουμε αυτές τις δύο πτυχές. Χθε αυτό είχα μια απόδειξη στην περιφέρειά μου συμμετείχα σε δύο διασκέψεις για ε, ανανεώσεις πηγές ενέργειας, για τη ρύθμιση των τιμών, ε, μιλούσαν για τις ανανεώσεις πηγές, ανανεώσεις πηγές ενέργειας, δίχως όμως να γνωρίζουν τις επιπτώσεις των βιοκαυσίμων. Ε, και πήγα και σε μια άλλη διάσκεψη του μια μη κυβερνική οργάνωση και έλεγε πώ η Ευρώπη έθεσε αυτό το 10% για το 2020 τα βιοκαύσιμα στις μεταφορές. Άρα λοιπόν έχουμε ανάγκη να δώσουμε μια μεγαλύτερη συνοχή στις επιλογές μας. Συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν από τους συναδέλφους και κρίνω ότι θα πρέπει να δείξουμε θάρρος εμείς Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι νομοθέτες, πως έχουμε στηρίξει και συνεχίζουμε να στηρίξουμε τον οδικό χάρτη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αρκεί να σκεφτούμε τι ψηφίσαμε προημερών στο, στην Ολομέλεια για το 2030 λέγοντας ότι έχουμε ε, κάνει κάποιο λάθος αν ε, θεωρούμε αυτό το 10% θα αντικαθίσει τα ε, κάψιμα τα ορυκτά από την ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εγώ, εγώ συμφωνώ ότι εδώ οι αγορές έχουν κάποιες προσδοκίες και θέλουμε θέλουν να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο έχουμε πει εμείς ως νομοθέτες και πρέπει να πούμε ότι επειδή σφάλαμε αυτός ο στόχος λοιπόν για την επικέντρωση στις συμβατικές μορφές εναλλακτικής ενέργειας και όχι στις πιο προωθημένες τεχνικά ίσως να υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι για να μειώσουμε τις εκπομπές και όχι μόνο η μείωση των, της χρήσης ορυκτών δεν κάναμε τις απαραίτητες ε, ε, μελέτες ε, εκτίμησης επιπτώσεων. Έχει, έχει δίκιο ο συνάδελφος. Οι επιπτώσεις δεν είναι αυτές που κρίναμε. Ε, αντίον θα είναι χειρότερες. Δηλαδή η αφαίρεση γεών από προϊόντα διατροφής και πόσα εκατομμύρια πληθυσμού θα τρεφόταν εάν αυτά τα εδάφη τα οποία έχουν, δοθεί στην παραγωγή βιοκαυσίμων θα είχαν φυσικά επιπτώσεις και για τις τιμές των πρώτων υλών των τροφίμων ε, και ίσως να μην είναι αυτές που έχουν εκτιμηθεί ε, και μετά το 2007 ξέρουμε ότι το αναγώσιτος της Αμερικανικής αγοράς είχε μια μεγάλη αύξηση λόγω των επιλογών που έκαναν. Λοιπόν, κατανοούμε αυτές τις επιπτώσεις και έχουμε την υποχρέωση να τις διορθώσουμε το πώς ε, υπάρχουν διαφορετικές λύσεις. Ε, κάποιοι λένε θα πρέπει να αφαιρέσουμε το όριο των 10% το μειώσουμε. Άλλος ε, έχει διαφορετική άποψη. Εγώ νομίζω θα βάλουμε, πρέπει να θέσουμε ένα ανώτατο όριο χαμηλότερο σαν αυτό της Κομισιόν είχε και ακόμα πιο χαμηλό, μιλάμε για 5% αλλά θα πρέπει να το εξετάσουμε. Θα πρέπει να κάνουμε ένα δικό χάρτη για την κατάργηση την ολική της χρήσης ε, υλών που θα μπορούν να είναι τροφικές ε, και να τις αντεκαταστήσουμε με προϊόντα πιο προηγμένα, αλλά και εδώ χωρίς να διαπράξουν τα σφάλματα που διαπράξαν αυτήν την οδηγία, διότι αν είναι να αντικαταστήσουμε αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις, τις συνέπειε διότι θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είναι απόρριμα κάτι το οποίο δεν είναι είναι, είναι ένα απόρριμα το οποίο μπορεί να πει στην γεωργία, δηλαδή κάποιο χρήσιμο υλικό. Όσοι λοιπόν κάνουν αυτές τις μελέτες αντικτύπου να τις κάνουν πολύ προσεκτικά ε, συνεργαζόμενοι με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, και να δουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από αυτές τις πολιτικές. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να διορθώσουμε την πορεία μας ε, και να εξηγήσουμε σε όσους υποστηρίζουν την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών διότι έχουμε κάνει κάποια σφάλματα, διότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ε, τόσο εύκολα και γρήγορα τις της πηγές ενέργειας και τελευταία παρατήρηση θα πρέπει να πούμε κάτι παραπάνω σχετικά με το e-look τώρα για τις έμεσες επιπτώσεις σχετικά με τη χρήση της γης θα πρέπει να υπολογιστεί μιλάμε για παρακολούθηση εποπτεία των επιπτώσεων αυτό δεν αρκεί νομίζω ότι όταν γίνονται οι παρακολουθήσεις αφού έχουν δημιουργηθεί προβλήματα δεν αρκεί πρέπει να το προ, προϋπολογίσουμε. Είμαστε προορατικοί λοιπόν σε ορυφάρε εκπομπέ και θα πρέπει να το ποσοτικοποιήσουμε. Είμαι βέβαιη πω η, Κομισιό, η Επιτροπή μα θα κάνει με πολύ καλή δουλειά και θα διορθώσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές σε κάποια ζητήματα. Μόνο οι ανόητοι δεν βλέπουν τις ε, αρνητικέ επιπτώσει των επιλογών του. Δεν άκουσα ο πλευρά παραγωγών ε, ε, επιχειρήματα πιστικά για να μην αλλάξει κάτι. Λέγεται πως ε, όλα τα κακά δεν αφορούν τα βιοκαύσιμα. Υπάρχουν και διαφορετικά διαφορετικές επιπτώσεις. Δεύτερον λέγεται να προστατεύσουμε τις επενδύσεις. Θεωρώ ότι μια προοδευτική πολιτική κατορθώνει να προστατεύσει τις επενδύσεις διότι μόλις ξεκινήσαμε στη χώρα μου π.χ. Ε, ε, ε, επικυρώθηκε δύο χρόνια πριν από δύο χρόνια αυτή η οδηγία άρα είμαστε στις αρχές και η προσπάθεια αντικατάστασης των ε, τροφίμων ε, με άλλες παραγωγές είναι διαθέσιμες ε, και θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τον χρόνο για να προσαρμοστούμε προς αυτές τις νέες επιλογές. Επαναλαμβάνω, ε, εγώ φοβούμαι ποια θα είναι η συνολική εκτίμηση και όχι η δουλειά αυτή κατά αυτή της Επιτροπής μας. Εμείς θα υποβάλουμε τις τροπολογίες μας τις προσεχείς ημέρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρινς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συντάκτη της γνωμοδότησης που παρουσίασε πολύ καλά τον προβληματισμό. Η Επιτροπή μας πρέπει να αναρωτηθεί περισσότερο για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε τους στόχους μας. Το δίλημα είναι ότι χρειαζόμαστε καύσιμα, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί να αφήσουμε τον κόσμο να πεινάει. Η οδηγία λοιπόν, αν εγκρίνονταν θα έλυνε το πρόβλημα. Αυτό είναι δηλαδή το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε. Κατά τη γνώμη μου μπορεί να συνεισφέρει σε κάποια λύση. Αλλά μην έχουμε ψευδεστήσεις. Αν η Ευρώπη απαγόρευε την εισαγωγή όλων των προϊόντων που ανταγωνίζονται τα τρόφιμα, θα είχε λυθεί το πρόβλημα. Ε, δεν νομίζω γιατί τότε θα αφήναμε το χώρο για άλλους. Γιατί δεν είμαστε οι μόνοι που είμαστε παρόντες στις υπονάπτυξη χώρες, για την αγορά δηλαδή ε, φυσικών πόρων. Προκειμένου λοιπόν να βρεθούν λύσεις πρέπει να επανέλθουμε στο βασικό. Και το βασικό είναι να μην είναι οι εταίροι μας. Πρέπει να δούμε μάλλον το κατά πόσο οι εταίροι μας έχουν ή δεν έχουν στα χέρια την υπόθεσή τους. Οι εταίροι μας δηλαδή στο Νότο μπορούν να αποφασίσουν όπως θέλουν. Γιατί εμείς λέμε ότι μπορούμε να ελευθερώσουμε ένα χώρο. Ποιος θα τον πάρει αυτό το χώρο. Η Κίνα είναι η πρώτη χώρα η οποία έχει καταλάβει ότι αρχίζουν να σπανίζουν οι πόροι και έχει αναπτύξει μια στρατηγική τέτοια που προσπαθεί να έχει εκείνη όλους τους πόρους. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσουμε λοιπόν τον αγώνα αυτό είναι να πείσουμε τους εταίρους μας στον Νότο να αναπτύξουν πολύ πιο ισχυρές στρατηγικές ώστε να διατηρήσουν τους πόρους τους και τους φυσικούς τους πόρους. Από εκεί απορρέουν μετά οι διάφορες επιλογές. Οπότε εγώ συμφωνώ με αυτό που είπαμε. Αλλά προσοχή μην είμαστε αφελείς και μην το κάνουμε απλώς ε, αυτομαστίγωμα. Ο πολιτικός διάλογος για να αξίζει το όνομά του πρέπει να πείσουμε τις χώρες του Νότου να υιοθετήσουν στρατηγικές τέτοιες που να φέρουν καρπούς στις ίδιες αυτές τις χώρες. Ό,τι άλλο έχουμε πει για την έμεση αλλαγή χρήσης γης, όλα αυτά πρέπει να εντάσσονται στον διάλογο για την Υπηρεσία εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφίβολα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα το λόγο, λέει Πρόεδρο, ο κύριο Όουεν. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και του άλλου ομιλητέ, για τις παρεμβάσεις του όπου εξήγησαν ε, τα θέματα που θεωρούν σημαντικά σε αυτό το πολύ πολύπλοκο θέμα. Είναι πολιτικό από τεχνική και από πολιτική άποψη. Υπάρχουν αρκετέ ε, επιτροπέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που το εξετάζουν και το Συμβούλιο το τελευταίο εξάμεινο εξετάζει το θέμα για να προσπαθήσει ε, να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του θέματος αυτού. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα από τα θέματα κλειδιά στην πρόταση της Κομισιόν είναι να μειώσει τις αντικές ε, συνέπειες ε, της έμεσης αλλαγής χρήσης της γης ε, και αυτό το κάνει με το ποσοστό του 5% όπου οι παραδοσιακές καλλιέργειες βιοκαυσίμων όπως είναι η τα κτλ. έχουν ανώτατο ποσοστό 5%. Έτσι προσπαθούμε να μειώσουμε τις εκπομπές που οφείλονται στην έμεση αλλαγή χρήσης της γης ενώ σεβόμαστε τις αποφάσεις σε οικονομικών φορέων να επενδύσουν στον τομέα αυτών ε, με τα κίνητρα που έδωσε η νομοθεσία τα τελευταία χρόνια. Ε, νομίζω ότι ήδη δηλαδή περιλαμβάνει η Κομισιόν ε, κάποια στοιχεία για ε, να μειώσει τις συνέπειε. συνέπειες. Ε, το άλλο θέμα είναι οι παράγοντε έμεις αλλαγής της χρήσης της ε, δηλαδή οι παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, ε, όταν υπολογίζουμε τις ε, εκπομπές που προέρχονται από την έμεση αλλαγή χρήσης της γης. Δεν λαμβάνονται λοιπόν υπόψη σήμερα οι παραγόντες αυτοί για να καθορίσουμε αν ένα βιοκάψιμο είναι βιώσιμο ή όχι. Θέλουμε όμως τα επόμενα χρόνια να συλλέξουμε τις πληροφορίες αυτές για να προγραμματίσουμε τι θα γίνει μετά το 2020 και να επικεντρωθούμε στα σωστά βιοκαύσιμα στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτό λοιπόν συνάδει με αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Η άλλη πτυχή που καλύπτει η πρόταση της Κομισιόν είναι το πώς ε, να χειριστούμε τα ε, ε, προηγμένα βιοκαύσιμα. Έχουμε κοιτάξει κάποια κάποιες καλλιέργειες που θεωρούμε ότι θα είναι οι καλλιέργειες του μέλλοντος. Προσπαθούμε Ε, να κοιτάξουμε και τα λοιπάσματα στο μέλλον ε, και τους τρόπους καλλιέργειας. Ε, και αυτό νομίζω ότι ακολουθεί αυτά που άκουσα σήμερα το πρωί. Πάντως η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να βοηθήσει οποιονδήποτε ευρωβουλευτή να καταλάβει τις τεχνικές στοιχές του φακέλου αυτού τις επόμενες εβδομάδες μέχρι την ψηφοφορία από ό,τι καταλαβαίνω, ε, η Ολομέλεια θα ψηφίσει αρχές σε Σεπτεμβρίου για το θέμα αυτό. Ε, στο μεταξύ θα ψηφίσουν οι επιτροπές. Ε, το θέμα πάντως είναι να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Υπάρχει πολλή αβεβαιότητα στον κόσμο σχετικά με το ποια είναι η πραγματική πολιτική μας, ποια είναι τα καλά βιοκαύσιμα, ποια είναι τα κακά βιοκαύσιμα, κάτι που καθυστερεί τις επενδύσεις αυτές αυτή τη στιγμή. Η Κομισιόν λοιπόν σίγουρα θέλει να συνεργαστεί με τα άλλα θεσμικά όργανα για να ε, διασφαλίσουμε την ολοκλήρωση του φακέλου αυτού ε, κατά την παρούσα θητεία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριο Κάσμαρετ ε, για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρετίζω τη συνένεση που προέκυψε ανάμεσά μας. Συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις που έγιναν σε ό,τι φορά την κυρία Τόγια Φυσικά δεν είμαι κατά της προστασίας των επενδύσεων, των αντίων. Είμαι υπέρ της προαγωγής αυτών, αλλά κάθε επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί στους, στα ζητήματα που εντάσσουν τις αρμοδιότητές της. Και η Επιτροπή ΙΝΤΕ δεν ασχολείται παραδείγματος χάρη με θέματα ανάπτυξης τρίτες χώρες, ασχολείται με τα θετικά πλονεκτήματα προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα σε έρχομαι τις έρευνες για το βιοκαύσιμα και τα προηγουμένα ιδιαίτερα πρόκειται να προωθήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι ουδής επιστήμων δεν μπορεί να μας εγγυθεί τα αποτελέσματα των μελλοντικών ερευνών. Μπορούμε φυσικά να προαγάγουμε τις έρευνες, αλλά δεν μπορούμε εκ των προτέρων να γνωρίζουμε κατά πόσο οι έρευνες αυτές θα έχουν θετικό αποτέλεσμα. Εάν η νέα γενιά βιοκαυσίμων θα είναι αποτελεσματική από οικονομική σκοπιά και κάτι ακόμα σχετικά με τα εδάφη, με τις γέες. Οργανώσαμε στη Ζιμπάμπουε μια συνάντηση, ήμουν παρόν μαζί με τον κύριο Νόησερ, ο οποίος το παρουσίασε την έκθεσή του στα, τον Ιούλιο εκεί. Εξετάσαμε ιδιαίτερα το ε, θέμα της ε, ε, ε, και της αναδιανομής των γεών. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξής. Πολλές γεές βρίσκονται για αγρανάπαυση δεν παράγουν ούτε τρόφιμα ούτε βιοκάψιμα. Ο πληθυσμός δεν έχει ακόμα τους, ε, τα στοιχεία σχετικά με την ιδιοκτησία των γεών αυτών, έχετε σχετικά έγγραφα θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και αυτού τους τίτλους ε, ιδιοκτησίας δίχως αυτούς τους τίτλους δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ούτε μηχανική παραγωγή ούτε ε, την ε, παραγωγή τροφίμων. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε πως αυτή η πολιτική θα είναι κατάλληλη. Τα νομικά ζητήματα έχουν μεγάλη σημασία και θα πρέπει να τα εξετάσουμε προσεκτικά. Ευχαριστώ. Υπενθυμίζω πως η κατάθεση τροπολογιών για αυτήν την έκθεση είναι 31 Μαΐου το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 24 Ιουνίου. Επιστώ την προσοχή σας ότι τώρα θα διακόψουμε την επιτροπή μας, τη συνάντηση και θα επανέλθουμε στις 15.00. Πρέπει παρακαλώ να είμαστε στην ώρα μας, διότι ο Επίτροπος Πίλμπακ θα έχει μόνο 30 λεπτά στη διάθεσή του. Θα πρέπει λοιπόν να επωφελθούμε κάθε λεπτού και άρα θα ξεκινήσουμε στις 14.59 ε, λεπτά. Ευχαριστώ.